Yes, I here on. Welcome. Good afternoon. Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι και καλό σας απόγευμα σας εύχομαι. Αρχίζουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων μετά την πολύ χρήσιμη ακρόση που είχαμε το πρωί για τον ανταγωνισμό. Καταρχήν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων 10 και 7 Μαρτίου και 22 Μαρτίου. Ωραία, εγκρίνονται. Ανακοινώσει του Προέδρου. Τρίτος ε, διάλογος ε, τριμερής έγινε για τον ΆΙΟΠ στις 13 ε, ημέρα Τρίτη. Αναφέρθηκαν πολλά θέματα, απαιτήσει πληροφοριών, η δήλωση ενδιαφέροντο και καλύπτουμε ένα φάσμα άρθρων. Καταλήξαμε συμβαστική λύση με μερικά μόνο κρεμή τεχνικά ζητήματα. Και πρόοδο σημειώσαμε και σε άλλα κέρια ζητήματα, όπως τα αποθετήρια και τις βασικές λειτουργίες. Ο επόμενος τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για την 4η Μαΐου. Περνούμε τώρα στο σημείο 5 κατεξουσιοδότηση κανονισμός επιτροπής για τη διόρθωση του κατεξουσιοδότηση κανονισμού 2015-63 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014-59 με θέμα τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης. έχει υποβληθεί επισήμω μια πρόταση αντίρρησης ή εναντίωση σε κατεξοδότηση πράξη που διορθώνει προηγούμενη κατεξοδότηση πράξη. Υπάρχει διάσταση απόψε ως προς την ερμηνεία της ένομης συνέπεια της νέας διορθωμένης κατεξοδότηση πράξης. Έχω λάβει επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΦΙΣΜΑ, του Ιράσεν, με ένα παράρτημα ερωταπαντήσεων. Ο Γενικός Διευθυντής μας παρουσιάζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί ότι ε, η νέα κατεξοδότηση πράξη δεν ε, διευρύνει το πεδίο εφαρμογή, απλώς κάνει μια ενημέρωση με κάποιες παραπομπές σε νομοθετικές διατάξεις που αναθεωρούν προηγουμένες και στις οποίες ε, αναφερόταν η αρχική κατεξοδότηση πράξη. Αυτή είναι η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι είναι τεχνική διόρθωση. Δηλαδή γίνεται απλώς ε, ε, διασταυρωμένη παράθεση και παραπομπή σε άλλες νομοθετικές διατάξεις. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ανησυχίες και ζήτησε διευκρινήσεις για το κατά πόσο όντως ισχύει αυτή η τεχνική απλώς διόρθωση ή μήπως κάποιες αναφορές, κυρίως στο άρθρο 429β προσθέτει κάποια στοιχεία. Επίσης υπάρχει ένα ερώτημα ως προς την αναδρομικότητα, του κατά πόσο ισχύει ή όχι. Έχουμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις και από τις απαντήσεις ε, θα καθοριστεί η περαιτέρω αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας δώσει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις και διευκρινήσεις. Θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουμε και την ενημέρωση που θα μας κάνετε, θα αποφασίσουμε τα επόμενα μας βήματα, μια και έχουμε ένα φάσμα επιλογών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον κύριο Εμιλιάνο Τορνέζε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, στην επιστολή μας στην επιστολή που σας έστειλε δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής μου προσπάθησε να σας εξηγήσει το σκεπτικό αυτής της διόρθωσης της κατεξοδότηση πράξης. Δύο βασικά είναι τα στοιχεία. Ε, ο κατεξοδότηση κανονισμός διορθώνει βασικά δύο σημεία που αφορούν την, ε, την, την αντιμετώπιση των τραπεζών πρόθεσης και επίση μία προσαρμογή ως προς τις αιτιολογικές σκέψεις σε ό,τι αφορά την ε, διασταυρωμένη παραπομπή στο CRR και κυρίως το άρθρο 429 που έχει αντικατασταθεί πλήρως. Η αλλαγή της αιτιολογικής σκέψης ε, δεν είναι σημαντική γιατί με βάση την κατεξοδότηση πράξη του 2015 ε, που τροποποίησε ε, το την προηγούμενη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία αυτή είχε αλλάξει από τον Ιανουάριο του 2015, οπότε ο διορθωτικός κανονισμός που δεν έχει εγκριθεί ακόμη, ουσιαστικά κάνει μια αυτή της αλλαγής χωρίς να τροποποιεί το ουσιαστικό δίκαιο από τον Ιανουάριο του 2015. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία του διορθωτικού κατεξοδότηση κανονισμού. Και όπως λέμε και στην οδηγία, αυτός ο διορθωτικός κανονισμός δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί η μεθοδολογία ε, άρχισε να ισχύει από τον Ιανουάριο του 2015. Επίσης δεν διεύρυνε το πεδίο εφαρμογή καν, που προσδιορίζεται από, την πρώτη από τον πρώτο κατεξοδότηση κανονισμό που αφορούσε τις συνεισφορές και αφορούσε ορισμένα μόνο παράγωγα και όχι το σύνολο των παραγωγών. Για παράδειγμα, το ισχύον 429 άρθρα παράγραφη 6 και 7 περιέχει αναφορά σε ε, δημιουργικά παράγωγα που δεν εμπίπτουν ε, στο πεδίο εφαρμογή ε, της ειδική αντιμετώπισης που απολαμβάνουν, της ειδική μεταχείρισης. Επίσης, η μεθοδολογία, επαναλαμβάνω, ισχύει από, την από τον Ιανουάριο του 2015, οπότε ο διορθωτικός κανονισμός δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα ή συνέπεια, ούτε πρόκειται να αλλάξει το ουσιαστικό δίκαιο που ίσχυε τότε. Ελπίζω να διευκρινίστηκε η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παρόλο που αντιλαμβάνομαι το ζήτημα είναι περίπλοκο. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χόκμαρκ, που είναι ο συντάκτης της αντίρρησης και θα ακολουθήσει συζήτηση. Ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ. Έχει απόλυτο δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προς την περιπλοκότητα του θέματος που είναι όντω πολύ σύνθετο. Φαίνεται ότι έχει δική του πορεία και ζωή αυτό το θέμα. Και εδώ και πολύ καιρό με την κυρία Φεραίρα θεωρούσαμε ότι είχαμε καταλήξει σε πολιτική συμφωνία. Και θεωρήσαμε ότι το ζήτημα Είχε λήξει όταν λάβαμε την καταξιοδότηση πράξη, αλλά τελικά πάλι εδώ είμαστε. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω έπρεπε να διορθώσει τον καταξιοδότηση κανονισμό εξαιτία των εξελίξεων που είχαμε στον κανονισμό κεφαλαικών απαιτήσεων. Βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, μπορεί να είναι σωστές ή αλλά υπάρχουν διστάμενες ε, ερμηνείες. Και μπορούμε να πούμε ότι προφανώς θα έχει συνέπεια και το πώς θα καταμετρήσουμε τις ε, πληρωμές στο Ταμείο. Θα εξαρτηθεί από την ερμηνεία που θα υιοθετήσουμε. Πάντως συνέπειες υπάρχουν. Και το κεντρικό ζήτημα εδώ είναι πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε το άρθρο 429 και την παραπομπή σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ενημερώνει, ε, επικαιροποιεί, διορθώνει κατεξοδότηση κανονισμό, κατά τη γνώμη μας διεύρυνε αυτή την παραπομπή, την αναφορά στο άρθρο, με την παραπομπή στο άρθρο 429. Εμείς θεωρούμε ότι με την αναφορά που κάνει στο άρθρο 329 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διόρθωση του κανονισμού διευρύνει και το πεδίο εφαρμογή. Το θέμα είναι πώς θα ορίσουμε αυτό το ευρύτερο πεδίο. Θα έχουμε κάποια επιρροή στα κονδύλια που θα καταβληθούν στο Ταμείο. Θα εξαρτηθεί αυτό από το αν η ερμηνεία μας είναι διασταλτική ή συσταλτική. Όταν είχαμε τη συζήτηση μεταξύ Σκεδόνης, Υγητών και επιτροπής, λάβαμε την άτυπη υπόσχεση ότι θα διορθωνόταν το πρόβλημα τη διόρθωση του διορθωμένου κανονισμού σε σχέση με τις παραπομπές που γινόταν στο 429α και β. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή γιατί δεν τήρησε την υπόσχεσή της, γιατί αυτό μας είχε υποσχεθεί και ότι θα γινόταν μάλιστα πολύ γρήγορα, μέσα στη, τη βδομάδα που μιλήσαμε. Και αυτή κατά τη γνώμη μας ήταν και η απλούστερη και ευκολότερη λύση. Και αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα χρειαζόταν καν να καθόμαστε εδώ πάλι και να συζητάμε το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ερωτώ λοιπόν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευρύνει την ερμηνεία της παρόλο που το διαψεύδει. Ενώ όλοι συμφωνούμε ότι δεν χρειάζονται όλες αυτές οι αναφορές στο α και β του 429. Είναι κάπως ομιχλώδη συζήτηση και πολύ περίπλοκη και σέβομαι αυτό το επιχείρημα ότι είναι περίπλοκο το θέμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε πλήρη ενάργεια και βεβαιότητα. Κατά τη γνώμη μου δεν το έχουμε υλοποιήσει. Θα το είχαμε καταφέρει αν είχε απαντήσει και αντιδράσει μέσα στη βδομάδα από τότε που είχαμε τη συζήτηση και την υπόσχεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Μάρκου Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Επειδή είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, όλοι συμφωνούμε ότι είναι περίπλοκο, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα που είναι πιο εύκολο για μένα. Εδώ τι πρόκειται. Πρόκειται για την κατανομή βαρών ε, του Ταμείου και δεν είναι τεχνικό, αλλά πολύ πολιτικό το θέμα. Σε τελευταία ανάλυση δηλαδή, ποιος πρέπει να συνεισφέρει πόσα στο ταμείο. Στο πλαίσιο της ε, νομοθεσίας, ε, αντικαθιστά εδώ το συνάδελφο Βόρτμαν Κόλ, στην αρχή των διαπραγματεύσεων λοιπόν καταπιαστήκαμε με το θέμα πώς τα net, οι διατάξεις netting μπορούν να εφαρμοστούν ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν εδώ. Και είχαμε συμφωνήσει ότι οι προϋποθέσεις netting δεν εφαρμόζονται στον υπολογισμό των συνεισφορών. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που ε, συζητήθηκε στο επίπεδο 1 και στο level 1. Στο level 2 δεν μπορεί να αλλάξει η θεώρηση. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, πόσο μάλλον που, υπάρχουν, ε, που θα ισχύσει και για τις συνεισφορές του 2015. Αν η Κομισιόν προτίθεται τη βούληση του, κοινοτικού, του ε, νομοθέτη του Κοινοβουλίου να την παρακάμψει, ε, αν θέλει να τη λάβει υπόψη, μπορεί να γίνει μέσω της ένστασης. Διότι η μπορεί να ε, συμπεριλάβει η Κομισιόν ε, τη διευκρίνηση που ζητεί ο κύριος Χέκμαρ, ότι δηλαδή η αναφορά περιορίζεται στο 429α ε, και όχι 429β και ότι αυτά δεν θα ισχύουν αναδρομικά αλλά από το 16 και μετά. Και θα πρέπει να υπάρχει και νομική βεβαιότητα σε όλα αυτά και νομική ασφάλεια γιατί οι ερωτήσεις-απαντήσεις που υπάρχουν υπάρχουν εδώ και καιρό στην ιστοσελίδα της Κομισιόν. Δεν διευκρινίζουν όμως αυτά που ζήτησα και εγώ μεταξύ άλλων στην επιστολή μου. Αν δεν γίνει αλλαγή, τροποποίηση με νομική ε, βεβαιότητα, τότε είναι σαν να καλούμε μέσω στις τράπεζες, μέσω της ίσπραξης των ε, συνεισφορών, να προσφεύγουν στα δικαστήρια και να αποφασίζουν τα δικαστήρια ε, ο σκοπός μας είναι, όπως είπα, η νομική ασφάλεια και όχι η νομική ανασφάλεια και η αβεβαιότητα. Γιατί η Κομισιόν δεν μπορεί πάνω στη βάση των όσων συζητήσαμε ήδη στα πλαίσια της διαπραγματευτικής ομάδας να προβεί σε τροποποιήσεις. Ε, θα ήταν εύκολο να λυθούν τα θέματα χωρίς μεγάλα προβλήματα και θα ε, ακολουθούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ ρωτώ λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα δεν κατάφερε η Κομισιόν να κάνει αυτές τις διευκρινήσεις που δεν ε, έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά στα πλαίσια των ερωτήσεων και απαντήσεων μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ε, ε έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι το λόγο, αλλά να είστε σύντομοι παρακαλώ έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Κανονικά έπρεπε να είχαμε περάσει στο επόμενο θέμα μας. Βεβαίως να συζητήσουμε, αλλά μη μακρηγορήσετε. Κύριος Μπάλτς, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ συνεχίζω μετά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Χόκμαρ και Φέρμπερ. Για μένα είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα να, να παραμείνουν διαφανή αν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις με αναδρομική ισχύ που είχε αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο, τότε και είχε τεθεί και σε ισχύ, δεν μιλάμε για διόρθωση της νομοθετικής πράξης, μιλάμε για, δεν μιλάμε για διόρθωση, μιλάμε για τροποποίηση της, νομο, της νομοθετικής πράξης. Και σωστά ζητεί το Κοινοβούλιο πρώτον να είναι διαφανής η διαδικασία και δεύτερον να υπάρχει και ε, πολιτική απόφαση που δεν θα αλλάζει με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν αλλάξει τίποτε σημαντικό, τότε νομίζω ότι θα πρέπει η Κομισιό να ξεκαθαρίσει, να μας διευκρινίσει εδώ ότι αυτό που συμφωνήσαμε ε, θα ισχύει στο τέλος. Η ε, επιστολή των υπηρεσιών της Κομισιόν αποτελούν διευκρινήσεις η διαδικασία των ερωταπαντήσεων ε, είναι μια ξεκάθαρη διευκρίνηση. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Γι' αυτό παρακαλώ και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια λύση η οποία θα σέβεται τις ε, νομοθετικές, τα νομοθετήματα που έχουν προηγηθεί και που θα φροντίζει και για την ύπαρξη νομικής ε, ασφάλειας. Ευχαριστώ, η Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι λίγο μπερδεμένη με τη σειρά των ομιλητών γιατί νόμιζα ότι οι σκιώδεις θα μιλούσαν αμέσω μετά τον κύριο Χόκμαρ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι στις 23 Φεβρουαρίου ε, που είχαμε τη συνάντηση με την Κομισιόν και ήταν ο κύριος Πάτρικ Πίρσον ε, και πάνω στη βάση εκείνη οι διευκρινήσεις δόθηκαν. Στις 17 Μαρτίου είχαμε την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έγγραφο με τις ερωταποκρίσεις που επιβεβαίωσε τα προλεχθέντα από τον κύριο Πάτρικ Πίρσον και ουσιαστικά νομίζω ότι ο στόχος του 1-2 του διορθωμένου κατεξουσιοδότηση κανονισμού έχει μια αναφορά που περιλαμβάνεται ε, στις ε, εκ των προτέρων συνεισφορές και το σχετικό κανονισμό για τη διόρθωση ε, σχετικά με το leverage ratio, το δίκτυ μόχλευσης. Συμφωνώ με την Κομισιόν εδώ. Το θέμα δεν είναι να επεκτείνουμε νομικά το πεδίο εφαρμογής των μέσων αυτών, το πεδίο εφαρμογή παραμένει καλά προσδιορισμένο και περιορίζεται από το άρθρο 5.3 αυτής της κρατεξουσιοδότηση πράξη και αναφέρεται στο παράρτημα 2 του κανονισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων. Δεν αλλάζει δηλαδή το εφαρμοστέο δίκαιο από τον Ιανουάριο του 2015 σε σχέση με την εκτίμηση των παραγόγων Υπάρχουν νέες διαπαραπομπές στο άρθρο 429, 429α, 429β του κανονισμού κεφαλαϊκών απαντήσεων του CRR δηλαδή, που ήδη είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Άρα δεν βλέπω λόγο εναντίωσης. Θεωρώ ότι είναι μια συγκλίνουσα ερμηνεία της νομοθετικής πράξης πάνω στην οποία εργαστήκαμε και σημειώνω επίσης ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην κατεξουσιοδότηση πράξη ε, παρά την κοινή δήλωση τη Γερμανίας, Αυστρίας, Ισπανίας και μια δήλωση της Σλοβενίας. Γενικά το Συμβούλιο συμφωνεί όμως. Ε, ειλικρινά μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε το θέμα. Δεν βλέπω δηλαδή λόγο ένστασης και εναντιόνσης. Ο κύριος Βεν Γίγκολτ. Πολύ σύντομα να πω ότι η συνάντηση των σχεδόν με την Κομισιόν ήταν από τις πιο αξιομνημόνευτες ε, συναντήσεις ε, σε πολλά επίπεδα. Γιατί φαίνεται παράδοξο, όπως έλεγε και ο εισηγητής, ε, ότι θεωρήθηκε και ισχυρίστηκαν ότι ήταν τεχνικό το θέμα. Μας υποσχέθηκαν εξηγήσει και μετά, όπως το έθεσε και ο Μάρκος Φέρμπερ, οι εξηγήσει που έφτασαν δεν έλυναν τα θέματα. Και αυτό συμβαίνει συνήθως όταν θέματα που ισχυρίζονται ότι είναι τεχνικά δεν είναι. Δεν συμφωνώ με την Ελίζα Φεραίρα λοιπόν. Εδώ υπάρχει μια ασυνέπεια. Στο άρθρο 1.3, όχι, στο 1.2 και μετά που άλλαξε το 5-3 της κατεξουσιοδότηση πράξη, γιατί λέει ότι πρέπει να περιορίζεται σε συμβάσεις παραγόγων αλλά μετά γίνεται αναφορά σε άρθρα τα οποία δεν αφορούν μόνο συμβάσεις παραγόγων και δεν μπορεί κανείς να μου εξηγήσει μέχρι τώρα και είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί η Κομισιόν δεν παρέδωσε τα υπεσχημένα γιατί δεν ε, ε, αρκεί να είμαστε στο 429α. Τότε θα είμαστε πολύ ευτυχείς όλοι, θα έλεγε η συζήτηση και θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν ανοίγει η πόρτα για περαιτέρω δυνατότητες netting που θα μετέθεταν τις συνεισφορές από τις μεγάλες τράπεζες που έχουν σημαντική έκθεση ως προς αυτό ε, σε μικρές τράπεζες. Ε, ενδεχομένως ε, η Κομισιόν θα έπρεπε να ε, ανταποκριθεί και να διευκρινίσει ότι είναι το 429α να σβήσουμε τις άλλες δύο αναφορές, τις παραπομπές και να πούμε ότι θα είναι ενιαία η έναρξη της εφαρμογής Πρώτου του 16. Και μετά, αφού κλείσει αυτό το θέμα, θα περάσουμε σε άλλα πιο ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, είναι σαφές. Υπάρχουν βέβαια ε, διστάμενες απόψεις, αλλά από τη δικιά μου τη σκοπιά έχω... υπάρχει μια ερώτηση που χρήζει απάντηση σαφέστερης. Η επιστολή του Γενικού Διευθυντού αναφέρει ότι η αλλαγή που αφορά την κατεξιοδότηση νομοθετική πράξη για το leverage ήδη είχε τεθεί, επειδή είναι δυναμική αυτή η παραπομπή. Οπότε η διόρθωση δεν είναι αμυγός νομική, μάλλον δεν είναι αμυγός απαραίτητη από νομική άποψη, γιατί λέτε ότι η νέα διάταξη με βάση τον κανονισμό για το leverage ε, τίθεται σε ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου του 2015. Είπατε ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ. Οπότε, η πρώτη ερώτηση που πρέπει να διευκρινιστεί. Αν όντω ισχύει αυτό, ότι δηλαδή ότι αυτό το συγκεκριμένο τμήμα που αλλάζει το νομικό, το νομικό θέμα, αλλά όχι και την ουσία, τότε γιατί κρίνεται σκόπι με τη διόρθωση αν η διάταξη, όπως είπατε, ήδη ισχύει από τον Ιανουάριο του 2015. Αυτά κατάλαβα εγώ από την επιστολή, εκτό και αν παρανόησα το περιεχόμενο της επιστολή. Δεύτερη ερώτηση. Για το 429β. Η αναφορά στο 429β είναι απόρρια του γεγονότο ότι για κάποιο τυπικό λόγο ε, ε, παραπέμψατε στο σύνολο του άρθρου, δηλαδή δεν είδατε ότι απαρτίζεται αυτό από τρεις παραγράφους. Αλλά γιατί αναφερθήκατε μόνο στο 429β και όχι μόνο στο α που θα προτιμούσαμε εμείς. Και το τρίτο ζήτημα αφορά την αναδρομικότητα. Είπατε ότι αυτό που ορίζει ο κατεξοδότηση κανονισμός είναι ήδη ενισχύ. Καταρχήν κατάλαβα καλά το περιεχόμενο της επιστολής. Ισχύει αυτό. Και επίσης τι με λιγενέστε τι βήματα πρόκειται να λάβει από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευκρινίσει περαιτέρω αυτά τα σημεία. Δηλαδή, από τις νομικές επιλογές που έχετε, ποια θα διαλέξετε για να κάνετε τη διευκρίνηση. Γιατί επί της ουσίας όλοι συμφωνούμε. Τώρα συζητούμε κατά πόσο υπάρχει αυτή η αφησιμία και πώς θα διαλευκανθεί. Πριν σας ξαναδώσω το λόγο για την απάντηση, ίσως ε, να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, του Ενίου Συμβουλίου Εξυγίασης και μετά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο Εξυγίασης έχει την ευθύνη για τις ε, ε, τράπεζες ε, στις 19 χώρες που συμμετέχουν στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Έχουμε συλλέξει τις σχετικές πληροφορίες για τις 762 τράπεζες που έχουν, στις οποίες έχει αποσταλεί η ενημέρωση ότι πρέπει να γίνει η συνεισφορά στον ενιαίο μηχανισμό, στο ενιαίο ταμείο στο SRF και έχουμε, ε, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία και επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Γιατί ήταν απαραίτητο να ενημερώσουμε τις τράπεζες με ξεκάθαρο τρόπο τι στοιχεία αναμέναμε από αυτές. Το ζήτημα είναι νομικό και ίσως να μην είναι προσφανοφρό αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε τις νομικές πτυχές του, αλλά από πρακτική άποψη ε, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, μάλλον να είναι ξεκάθαρο στις τράπεζες, ότι μόνο τα παράγωγα καλύπτονται από το άρθρο 429α για παράδειγμα τα παράγωγα χρεογράφων Ζητήσαμε από τις τράπεζες να μην τα λάβουν υπόψη τους ούτε ασφάλιστα. τα οποία καλύπτονται από το 429β. Και αυτό γιατί ο κανονισμός 63 ε, ε, του 2013 δεν τους το επιτρέπει. Είναι γνωστό ότι εμείς δεν συμμετείχαμε στις ε, συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων, το Κοινοβουλίο και της Επιτροπής επί του θέματος, αλλά εμείς η πρακτική συμβουλή που στείλαμε στις τράπεζες είναι να κάνουν της, ε, ε, επανεκτίμηση της αξίας μόνο των παραγόγων, γιατί μόνο αυτά θεωρούμε ότι καλύπτονται από το 329α. Ευχαριστούμε, η Επιτροπή. Το ζήτημα δεν είναι μόνο περίπλοκο από τεχνικής απόψεως, μιας και αφορά στα παράγωγα, αλλά επίσης και από νομοθετικής απόψεως. Και αυτό είναι ο λόγος που χρειαστήκαμε τόσο πολύ χρόνο για να αξιολογήσουμε τις πιθανές ε, λύσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ένα από τα ερωτήματα που θέτεται είναι εάν μπορεί να υπάρχει διόρθωση της διορθώσεως. Και η απάντηση είναι πως όχι, γιατί εδώ δεν υπάρχει ένα λάθος ε, τα πραγματικά περιστατικά, στα στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο και είναι αυτό κάτι που δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Την πράξη την υιοθέτησε το Συμβούλιο των Επιτρόπων, επομένως το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια διόρθωση σε αυτήν, δεν μπορεί να γίνει μια διόρθωση στην, στον διορθωτικό κανονισμό. Επομένως, για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια, όπως αναφέρθηκε, η Επιτροπή οργάνωσε workshop, στα οποία κάλεσε εκπροσώπους κρατών μελών και το Κοινοβούλιο, δια τη γραμματείας του, ε, όπου ζητήθηκε, ακούστηκε ότι πρέπει να ξεκαρθαριστεί η μεθοδολογία. Το Δεκέμβριο του 2014 μάλιστα δημοσιεύθηκαν και οι σχετικές ε, ε, ε, ερωτήσεις και απαντήσεις που έδιναν αυτή την κατεύθυνση. Πολύ δηλαδή πριν την υιοθέτηση του πρώτου διορθωτικού. Τις ίδιες απαντήσεις δώσαμε και σε άλλες περιπτώσεις όσον αφορά για παράδειγμα τις προθετικές ενέργειες των τραπεζών. Θέλαμε για λόγους αποτελεσματικότητας να έχουμε εγκρίνει μία πράξη, όχι δύο, αλλά τα κράτη-μέλη μας εφέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι αυτό ίσως δημιουργήσει σύγχυση. θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης γιατί ήδη εφαρμόζεται ουσιαστικά αυτή η νομοθετική πρόνοια, αλλά εν τέλει αποφασίσαμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί. Εξετάσαμε επίσης το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί μια πράξη η οποία να μεταθέτει την ημερομηνία εφαρμογή αυτού του κανονισμού την 1η του 2016. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει επειδή θα ήταν μεταβολή αναδρομική του ουσιαστικού ε, περιεχομένου της νομοθεσίας. και Και αυτά τα στοιχεία λοιπόν ελήφθησαν υπόψη στην μελέτη που συνόδευε την κατεξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής. Και γι' αυτό υπάρχει μια συγκεκριμένη ασφαλιστική δικλίδα. Για να περιοριστεί το επιτρεπόμενο netting των ε, παραγωγών, το επιτρεπόμενο συμψηφισμός. Στι αναφορέ του 329α και β ακολουθήσαμε την ίδια τεχνική με, τις με τον προηγούμενο κανόνα ε, πράξη. όπου δηλαδή γίνεται σαφής αναφορά σε credit derivative, σε πιστοτικά παράγωγα. παρά το γεγονός ότι τα πιστοτικά παράγοντα αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί το πεδίο εφαρμογή στον κανονισμό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αναφέρεται σε παράγωγα που καλύπτονται στο, παρά... του κανονισμού κεφαλαϊκής... ε... κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Έχω και μια τεχνική ερώτηση. Γιατί πολύ σωστό το επιχείρημα ότι ο προηγούμενος κατεξοδότηση κανονισμός αναφέρθηκε κατά δύο παραγράφους 6 και 7 του 429 που ενσωματώνουν και αναφορές σε άλλα ε, νομοθετικά μέσα που δεν καλύπτονται. Θα μπορούσατε όμως από ότι σε αυτήν την περίπτωση ε, παραθέσατε συγκεκριμένη παράγραφο και όχι το σύνολο το άρθρο. Γιατί στον, στο νέο κανονισμό έχει, αναφέρετε ολόκληρο το άρθρο που έχει όμως τρία μέρη και επικεντρώνεστε σε ένα μόνο μέρος. Γιατί αυτό ήταν αναπόφευκτο, γιατί στην ίδια παράγραφο έπρεπε να κάνατε την παραπομπή και στην περίπτωση αυτή αποφασίσετε να τα συνοψίσετε. Γιατί, γιατί αυτή η αλλαγή. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ακριβώς η ίδια η κατάσταση, υπάρχει διαφορά. Μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος. Όπως είπα, η νέα κατεξιοδότηση πράξη που προβλέπει αυτό το leverage ratio αντικαθιστά το 429 και αναφέρεται μόνο στο 429, 429α και 429β ως προς τη μεθοδολογία. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αυτή η μεθοδολογία δεν καλύπτει και άλλα νομοθετικά μέσα που δεν καλύπτονται από την νομοθετική πράξη. Αυτό είναι σαφές. Για παράδειγμα, το ενιαίο Συμβούλιο Εξηγήσεις δεν το εφαρμόζει και σε άλλα μέσα που δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Οπότε δεν υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει λάθος, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε πλέον τον κανονισμό τροποποίησης. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μάρκου, σύντομα. Δύο, δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, όταν ως Κοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουμε τη δυνατότητα να παραπέμπουμε κατά πράκτης, πράξης, ε, δεν ε, μπορούμε να βασιζόμαστε στο ότι ε, αν η μία ξεκινήσει τη διαδικασία θα συμφωνήσει η άλλη και οι δύο πρέπει να συμφωνήσουν εμείς δηλαδή θα πρέπει να ελέγξουμε αν θα συμφωνήσουμε ή αν θα απορρίψουμε την πρόταση αυτή. Η Κομισιόν έχει το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας. Πριν δηλαδή μπλεχτούμε σε νομικές διαδικασίες τι γίνεται και τι δεν γίνεται, το απλούστερο είναι να αποσύρει η Κομισιόν την πρότασή της και να υποβάλει καινούρια για να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου. Γιατί ε, δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει γιατί δεν αποσύρει την πρόταση να υποβάλει μια νέα. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είπε ότι είναι σαφές ότι ισχύει μόνο για τα παράγωγα. Και ούτως ή άλλως ίσχυε και από πριν. Οπότε αν ισχύει ήδη και από πριν, τότε ποια είναι η συνέπεια σε περίπτωση απόρριψης. Πέραν το ότι άλλες ε, διατάξεις θα καταπέσουν. Ποιο θα ήταν η ένομη συνέπεια αν δεν τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθετική πράξη. Δεν ξέρω βέβαια τι σχετισμό δυνάμεων υπάρχει να ψηφίσουμε, αλλά με ενδιαφέρει αυτή η πιθανότητα. Όπω είπα, το μόνο ουσιαστικό τμήμα τη κατεξοδότηση πράξη αφορά τι ε, ενδιάμεσε τράπεζε και τι τράπεζε προώθηση. Και αντίρρηση ένσταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για αυτέ τι τράπεζε. Σε ό,τι αφορά τα παράγωγα, ισχύει ήδη ε, νομοθεσία. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε διορθωτικό επιπλέον στον κανονισμό διόρθωση. Μάλιστα. Τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία. Είναι σαφές ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς την ερμηνεία. Δεν πρόκειται να λάβουμε απόφαση, απλώς ήταν ευκαιρία για να ακούσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, υιοθετούμε διαφορετικές ερμηνείες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το παράδοξο είναι ότι αν ε, υπερψηφιστεί η αντίρρηση, δεν θα επηρεάσει την αλλαγή. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο σχετισμό μεταξύ του αιτήματο ε, αντίρρησης και της ε, ένσταση ως προς τη διευκρίνηση. Και αυτό είναι, αυτή είναι και η πρωτοτυπία του μηχανισμού αυτού. Αλλά είναι και τμήμα της περιπλοκότητας της δημοκρατίας. Εν ναι, αυτό το χρόνο θα λάβουμε και απόφαση ως κυρίαρχο θεσμικό όργανο, αν ζητηθεί και ψηφοφορία, θα γίνει. Γκόναρ, αν δεν έχεις κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό να πεις, ουσιώδες, υπάρχει διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και θεωρίας. Υπερισχύει η πραγματικότητα. Αν καταλήξουμε συμφωνία, ποια θα είναι η βάση για τη συνεισφορά. Γιατί αν δεν υπάρχει ασάφεια στα έγγραφα, αν δεν υπάρχει σαφήνεια στα έγγραφα, αν υπάρχει ασάφεια, τότε ε, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει αυτή τη σαφήνεια. Αν δεν μπορεί να διορθώσει περαιτέρω τον κανονισμό της διόρθωσης, βρει άλλο τρόπο. είναι φαίνεται στο Q&A, αλλά κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποκαταστήσει τη σαφήνεια και την ασφάλεια δικαίου. Γιατί ως προς τη βάση συμφωνούμε. Δεν είναι εκεί που έχουμε διαφωνία. Το θέμα είναι η ερμηνεία. Θα πρέπει να θετήσουμε ίδια ερμηνεία. Κάποιος τρόπος θα βρεθεί. Και αυτό είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλει μαγεία πια για κάτι τέτοιο γιατί είναι δύσκολο να συζητούμε πάντα τόσο περίπλοκες ε, λεπτομέρειες. Πολύ σοφά τα λόγια σου, Γκούνερ. Αν μη τι άλλο, συμφωνούμε τη επί της ουσίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε η συγκεκριμένη ε, διάταξη να ε, εφαρμοστεί. Το netting μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία παραγόγων. Το θέμα είναι, θα είναι αυτό το αποτέλεσμα του κανονισμού. Αλλά το γεγονό ότι όλοι έχουμε το, τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό, αυτό είναι πολύ θετικό. Το θέμα είναι, είναι αρκετά σαφέ το κείμενο ώστε να ελοποιηθεί ο κοινό μα στόχο. Και έχει δίκιο ο Γκούναρ ότι υπάρχουν διάφορε επιλογέ και μεταξύ του να μην γίνει τίποτα και να διορθωθεί περαιτέρω διορθωμένος κανονισμός, υπάρχει και κάποια ενδιάμεση λύση. Και αν από τις ερωταπαντήσεις ε, δεν προέκυψε σαφήνεια, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί και να αποκαταστήσει τη σαφήνεια σε ένα θέμα που είναι προφανώς τεχνικό, δεν είναι θέμα ερμηνείας του δικαίου, γιατί όλοι θέλουμε η συγκεκριμένη διάταξη να τεθεί σε ισχύ. Ως προς αυτό συμφωνούμε, υπάρχει σύμνοια. Οπότε Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια θα τη συζητήσουμε με την κανονική διαδικασία. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίασης για την ενημέρωση και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μια στιγμή να βρω ποιο είναι. Το σημείο 6, τα εικονικά νομίσματα Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της έκθεσης του Γιάκοπ Φον Βάιτσέκερ. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ...128 τροπολογίες κατατέθηκαν... ...που είναι αρκετά λογικός αριθμός αντιμετωπίζεται... Και τις τελευταίες εβδομάδες, και αυτό είναι καλό, επιτελέσαμε σημαντική πρόοδο συμφωνώντας σε συμβιβαστικές τροπολογίες με βάση τις 128 κατατεθήσεις. Και κρίνοντας από μια συνάντηση που μόλις έλαβε χώρα μεταξύ Σιγητού και Σκιωδών σήμερα το απόγευμα, νομίζω ότι θα μπορούμε να πάμε ε, στην ψηφοφορία σύμφωνα με το πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα. Ακόμα δεν τελειώσαμε τα πάντα, υπάρχουν ορισμένα εκκρεμή, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις τροπολογίες που θα βελτιώσουν το κείμενο. Είχαμε καλές συζητήσεις, καλούς εμπειρογνώμονες και πολύ χρήσιμη συμβολή από το, τη γραμματεία και τους συνεργάτες μας. Η βασική ιδέα της έκθεσης πρωτοβουλίας νομίζω ότι παραμένει αμετάβλητη. Η ιδέα είναι ότι εδώ έχουμε μια νέα και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία η οποία εξελίσσεται ακόμα τόσο ραγδαία που δεν θα ήταν καλό να καταπνίξουμε την καινοτομία ε, προχωρώντας σε ρύθμιση εκτενή τώρα. Ενδεχομένως αυτό ενέχει κάποιους συστημικούς κινδύνους. Η χρήση θα γίνει σημαντική και αντί για νομοθεσία προφύλαξης προληπτική θα χρειαστούμε παρακολούθηση προληπτική προφύλαξης ε, και ούτως ώστε αν παραστεί ανάγκη να προχωρήσουμε σε νομοθετικά μέτρα γρήγορα πριν συμβεί κάτι άσχημο. Ένας τρόπος να το διατυπώσουμε αυτό είναι να πούμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε μία προσέγγιση πειραματική. Θα τα δοκιμάσουμε όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να ε, φτιάξουμε ε, έναν ε, ουρανοξύστη πάνω σε αμμώδες έδαφος. Ακόμα το έδαφος είναι αμμώδες. πριν προχωρήσουμε σε οικοδόμημα θα πρέπει τα θεμέλια να είναι στερεά. και σε αυτά τα πλαίσια θα βρούμε και συμβαστικές λύσεις. Θέλω να αναφέρω ιδιαίτερα δύο σειρές ε, τροπολογιών από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες συναδέλφους που αφορούν τη χρήση του DLT για την βελτίωση των εθνικών κτηματολογίων. Αυτό δείχνει τις ευρείες δυνητικές εφαρμογές της, κατανεμημένης, ε, της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και τις τροπολογίες 84 με 86 Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ χρήσιμη αναλογία μεταξύ της εξέλιξης του διαδικτύου και του ενδεχόμενου ε, δυναμικού που θα έχουν αυτές οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση επί των τροπολογιών ευρύ, ε, περισσότερο σε αυτή την ευρύτερη ομάδα. Όπως είπα όμως έχουν προχωρήσει πολύ οι εσωτερικές συζητήσεις και θα μπορούσαμε ε, να κυκλοφορήσουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών πολύ πριν από τη, μέρα της ψηφοφορίας για να προετοιμαστείτε όλοι ανάλογα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μαρτουσέλο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Γιάκομπ, ε, τον εισηγητή. Να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους σκιώδης που εργάστηκαν σε αυτό το φάκελο. Οι εργασίες προχώρησαν πολύ ικανοποιητικά. Καταλήξαμε στα περισσότερα θέματα και οι μεγαλύτερε ομάδε ε, ψηφίζουν υπέρ των συμβιβαστικών. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με τη δημιουργία μιας task force, μιας ειδική ομάδας, ε, για να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Γιατί τα κόστη είναι ασαφή και η επάντρωση είναι επίσης ε, ασαφής. πρέπει τα καθήκοντα μιας τέτοια ομάδας να είναι πολύ σαφέστερα προσδιορισμένα. Και αμφιβάλλω για το αν χρειάζεται πρόθεσμα νομοθεσία, γιατί η συζήτηση για τα εικονικά νομίσματα είναι μόλις στην αρχή της. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του εισηγητή. Ε, ε, είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα που θα βρίσκει σύμφωνα στις περισσότερες ομάδες και τη δική μου. Το εισηγητή ε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά προσπαθώντας να συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις. Ashley Fox. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις για το έργο τους ως τώρα, ιδιαίτερα τον Ιάκοπ για το εξαιρετικό έργο που έχει ε, καταβάλει για να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Οι κυριότερες ανησυχίες μας ε, της πολιτικής μου ομάδας είναι το κατά πόσον θα μπορούσε να επεκταθεί η οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπνήματος ξεπλήματος μαύρου χρήματο για να καλύπτει και τέτοιου τύπου συναλλαγές και η δημιουργία της ομάδας ε, εργασίας του Task Force. Όσον αφορά αυτήν την ομάδα εργασίας του Task Force. Είμαστε πλέον ικανοποιημένοι γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, κρατών μελών για να επεξεργαστούν νομοθεσία για αυτού του είδους τα εικονικά νομίσματα και τα τεχνολογία καταναλωμένου καθολικού. Γνωρίζουμε ότι τέτοια νομοθεσία δεν υπάρχει. Και επίσης συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών που θα μπορέσουν να μας δώσουν ε, τις πληροφορίες και να εξετάσουν τις εξελίξεις. Δεν θέλουμε με την ομοθεσία να πάψει να υφίσταται αυτή η τεχνολογία. Και με αυτή την θέση συμφωνεί και ο εισηγητής. Επομένως, συμφωνούμε ότι η πιθανότητα να υπάρξει ρύθμιση και νομοθεσία είναι μόνον εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι πρόσφορο για να μην υπάρξει κατάχρηση των εικονικών ε, νομισμάτων και αυτής της τεχνολογίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις για όλα τα ανοιχτά ζητήματα και οι συνάδελφοί μου συνεχίζουμε, και εγώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε για την Άλντε, ο κύριος Πιεταριάτσικ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την ε, επικοδομητική ε, στάση που έχει κρατήσει στις συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές και το έργο του και χαίρομαι που έχει αποδεχθεί πολλές από τις προτάσεις ε, και τροπολογίες που κατατέθησαν. Καταφέραμε μάλιστα σήμερα στη συνάντηση των σκιωδών να προχωρήσουμε πολύ όσον αφορά τα, τις συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ προσπάθησα να ξεκινήσω από τις ιδέες του εισηγητή και να τις αναπτύξω περισσότερο. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες έχουν και πολλά πιθανά ωφέλη τεχνολογίε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού μπορούν να ε, μειώσουν το κόστο συναλλαγών, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του εμπορίου μέσω ίντερνετ, μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ε, για παράδειγμα στη φορολόγηση και να βοηθήσουν ακόμα και τι δημόσιες αρχέ στο υποπτικό του έργο. Αλλά υπάρχει η πιθανότητα και το εικονικό νόμισμα να χρησιμοποιηθεί ε, με δυσμενεί επιπτώσει, με προβλημογόντας προβλήματα, καταχρώμενοι οι χρήστες του την ανωνυμία, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι χρησιμοποιείται το εικονικό νόμισμα για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών, για παράδειγμα. Αλλά είναι ένας κίνδυνος, τον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε στην έκθεση. Και όσον αφορά την ομάδα εργασίας, το Task Force, θεωρούμε ότι ε, είναι ορθό να δημιουργηθεί μια τέτοια ομάδα υπό την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε προτείνει κάποιες τροπολογίες που αφορούν στην εντολή της και στην σύνθεσή της. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα αυτή θα λειτουργήσει ως μια ομάδα παρακολούθησης η οποία θα φροντίζει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, ποιες είναι οι εξελίξεις, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση, εάν χρειαστεί, να υιοθετήσουμε νομοθετικά και πρωτοβουλίες και να ρυθμίσουμε τον τομέα αυτό. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτομάτως ξεκινάμε μια ρύθμιση. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ τώρα, της Ανατικής Αριστεράς, ο κύριος Μιγέλ Βιέγας. Εδώ μιλούμε για μια νέα τεχνολογία με τεράστιο δυναμικό ο φόβος μας είναι μέχρι ποιο βαθμό ε, θα ήταν πρώιμη μια πιθανή νομοθετική ρύθμιση. Μήπως μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση θα δώσει ένα σφαλμένο μήνυμα ε, καθησυχασμού σε μια τεχνολογία που αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα που θα πρέπει να επιλύσει στο μέλλον, γιατί βρίσκεται στα σπάργανα ακόμη. Και πολλά ερωτηματικά απομένουν ανεπίλητα δεν γνωρίζουμε καν ποιες θα είναι οι βασικές ε, λειτουργίες ε, των νομισμάτων με βάση τη νέα τεχνολογία. Είναι πολύ ευαίσθητα όλα αυτά τα σημεία. Και από τη στιγμή που οι εξελίξεις είναι ραχδαίες και τα εικονικά νομίσματα εξυπηρετούν ε, τα συμφέροντα μεγάλων χρηματοοικονομικών ομάδων, μήπως θα πρέπει να κάνουμε μελέτες και να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες τις εξελίξεις. Και μία ε, σφαιρική προσέγγιση θα πρέπει να ανταποκρίνεται ε, στις επιθυμίες όλων των πολιτικών ομάδων και αυτή την άποψη νομίζω τα κατάφερε ο εισηγητής. Υπάρχει ένα μεθοδολογικό ζήτημα, το, το κόστος των συναλλαγών, των συνδιαλλαγών. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι ε, σε τι περιορίζονται ε, αυτά τα κόστη. Όταν λέμε κόστος συνδιαλλαγής δεν είναι μόνο ε, ένα περιορισμένο κόστος. Έχουμε την αβεβαιότητα και ένα σύνολο στοιχείων που δεν περιορίζονται στα αμυγός τεχνικά σκέλη της συνδιαλλαγής. Γιατί εγώ μπορώ να αγοράσω σε ευτελή τιμή ένα προϊόν που κοστίζει φτηνά στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος συνδιαλλαγής είναι μηδενικό, γιατί στο κόστος συνδιαλλαγής υπησέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες, ε, τις πληροφορίες, ε, ενημέρωση και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα, πάντως ε, η τελική λύση μου φαίνεται καλή και δεόντως περιεκτική. Σας ευχαριστώ Μιγγέλ. Για τους πράσινους τώρα, το λόγο η κυρία Μόλι Σκοτ Κάτω. ήταν πολύ ε, χρήσιμη αυτή και με ικανοποίησε πολύ αυτή η ενασχόληση με το θέμα. Μου θύμισε τα χρόνια μου από το Πανεπιστήμιο. Είχαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια με εμπειρογνώμονες. Μάθαμε πολλά και ελπίζουμε ότι ε, κάναμε καλό έργο στο Κοινοβούλιο με τις τεχνολογίες του blockchain, της αλυσίδας επιβεβαιωμένων ομάδων συναλλαγών και πολύ συνεργάσιμο το όλο κλίμα. Πρώτη φορά σε ε, τέτοια διαδικασία είχαμε τόση συμφωνία και μεγάλη σημεία επί των συμβαστικών λύσεων. Εμείς ε, είμαστε υπέρ της ιδέας των εναλλακτικών νομισμάτων και είμαστε και υπέρ των τοπικών, περιφερειακών νομισμάτων που δίνουν ε, διεξόδου στην τοπική οικονομία. Μερικές φορές είναι εικονικά και άλλες φορές είναι... Ε, είναι, έχουν υλικό ε, υπόθεμα. Πάντως σχετίζονται κυρίως με ήδη, ένα συγκεκριμένο είδος συναλλαγών και δεν είναι και ανταλλάξιμα πάντα. Πάντως, οποιοδήποτε νομοθετική πρόταση που θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει, να φημώνει τις δυνατότητες αυτών των εικονικών νομισμάτων. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που σε αυτό το θέμα συμφωνήσαμε και με τον Άσλι Φόξ, που παρόλο που είμαστε συμπατριώτες, πολύ συχνά διαφωνούμε για πολλά θέματα. Αλλά εδώ συμφωνήσαμε. Ε, το θέμα της ε, κατανάλωσης ενέργειας ε, που είναι συναφής με τα εικονικά νομίσματα, γιατί διαπίστωσα ότι είναι μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ε, σε ό,τι αφορά την διανομή αυτή της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Θα πρέπει να βρούμε πιο φιλικέ προ το περιβάλλον λύσει. Γιατί βέβαια η ενεργειακή κατανάλωση λαμβάνει χώρα αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μα αφορά. Και μάλιστα από μια επιστημονική επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου διαπιστώσαμε ότι μόνο από το bitcoin έχουμε ένα γιγαμπάι το χρόνο ενεργειακή κατανάλωση. Είναι αντίστοιχο με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματο ε, ολόκληρη τη Ιρλανδία για ένα χρόνο. Οπότε αυτό το θέμα τη ενεργειακή κατανάλωση είναι σημαντικό. Μάλιστα θα εκπονήσουμε και σχετική τροπολογία γιατί μας προβληματίζει και νομίζω ότι περιλαμβάνεται και στις συμβαστικές τροπολογίες. Επίσης το θέμα των παραγόγων που σχετίζονται με τα εικονικά νομίσματα. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τη φύση τους και μετά να επεκταθούμε στα παράγωγα. Άλλο θέμα. Θέλουμε σωστό ορισμό για το ε, θέμα των χαρακτηριστικών του εικονικού νομίσματος και το θέμα της ανωνυμίας. Ε, προσοχή, γιατί μπορεί να έχουμε παράνομα προϊόντα, υπηρεσίες, χρηματοδότηση τρομοκρατία ή και φοροαποφυγή που να ενισχύεται από την εκτεταμένη χρήση αυτών των οικονομικών νομισμάτων. Είμαστε υπέρ της καινοτομία, αλλά να μην ξεχνούμε και του κινδύνου που ενδεχομένω ελοχεύουν με την χρήση τέτοιων νομισμάτων. Ο Μάρκο Τζάνι από το EFTD. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του, να συγχαρώ και τους βοηθούς του, αλλά και τους συναδέλφους, γιατί το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική βάση για να ξεκινήσουμε πιο συγκεκριμένες συζητήσεις ε, και κανονιστικού χαρακτήρα για τέτοιου είδους ε, μέσα που είναι τα εικονικά νομίσματα. Πολύ σωστά λέει η έκθεση ότι τα εικονικά νομίσματα έχουν τεράστιο δυναμικό, ιδιαίτερα σε δύο τομείς, ε, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και ε, την ανάγκη μιας φορολογικής διαφάνειας. Είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και τα εξετάζουμε και διεξοδικά και εμβριθώς. Επίσης ε, υπάρχει η δυνατότητα ενός εναλλακτικού και ανταγωνιστικού συστήματος πληρωμών από αυτό που διαχειρίζονται σήμερα οι ιδιωτικές τράπεζες. Οπότε πολύ σημαντικό το δυναμικό των εικονικών νομισμάτων. Αλλά υπάρχουν και δυνητικοί κίνδυνοι που θα πρέπει ε, να ληφθούν υπόψη και αυτό το αναφέρει πολύ εύστοχα ο εισηγητής. Επαναλαμβάνω, ως προς το κείμενο είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και μπορεί να έχουν απομείνει κάποιες λεπτομέρειες για την ομάδα εργασίας, την ειδική ομάδα κρούσης που προτείνεται, αλλά νομίζω ότι και αυτές τις μικροδιαφωνίες θα τις εξαλείψουμε στο τέλος, ώστε το τελικό κείμενο να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μπάρμπαρα Κάπουλ, τελευταία εκ των σχεδόν. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ιδιαίτερα για, τις, για τους πολύ ενδιαφέροντες γύρους συζητήσεων με τους ειδικού. Πράγματι θύμιζε πανεπιστήμιο και μάθαμε πολλά για την τεχνολογία της αλυσίδας των μπλοκ, του κατανεμημένου καθολικού κλπ. Και βρήκαμε και καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες στην τελευταία ιδιαίτερα σήμερα το μεσημέρι. Και η βασική ιδέα που με βρίσκει σύμφωνη και την είπε ο εισηγητής είναι οι καινούριε πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες που δεν πρέπει να φρεναριστούν ε, και αντιμετωπίζονται καλά από τον εισηγητή. Ε, προτείνεται μια ανάλογη ρυθμιστική προσέγγιση για να μην δημιουργήσουμε προσκόμματα. Το κόστος πρέπει να παραμείνει χαμηλό και οι ρυθμιστικές προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάλογα με τις εξελίξεις. Ε, βέβαια τα εικονικά νομίσματα συνεπάγονται και κάποιο ρίσκο στον τομέα της μαύρης αγοράς, της φοροαποφυγής, ε, του ξεπλήματος χρήματος και προφανώς όλα αυτά θα πρέπει να μπορούν να διώκονται η ψευδονυμία, η χαμηλή, η χνηλασιμότητα ε, κάποιων συναλλαγών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης αναφέρεται ότι η φυστάμενη νομοθεσία στην Ένωση, αυτή θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται. Το πιο σημαντικό όμως είναι να υπάρχει και εξατομικευμένη νομοθεσία για τα εικονικά νομίσματα. Ανάλογα με τα ε, αιτήματα των κρατών μελών, ε, καλύπτονται και οι πλατφόρμες που αφορούν τα εικονικά νομίσματα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ε, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός για τα εικονικά νομίσματα. Θεωρούνται ως ψηφιακή ε, αναπαράσταση μιας τιμής ε, που χρησιμοποιείται από μια αρχή. Τα εικονικά νομίσματα γίνονται δεκτά ως μέσα πληρωμών και μπορούν να καταγράφονται και να αποθηκεύονται. Γίνεται και μία εκτενής ανάλυση των εικονικών νομισμάτων για τη βελτίωση του ανταγωνισμού, για τη μείωση του κόστους των συναλλαγών. Πρέπει να γίνουν και stress test. Πολύ σημαντικό είναι το μεγάλο δυναμικό εξάπλωση των ψηφιακών τεχνολογιών και των εικονικών νομισμάτων. Θα πρέπει ε, που ξεπερνάει τον ε, ε, χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτό ελήφθη υπόψη από την εισήγηση που έλαβε υπόψη πολλές εφαρμογές που προβλέπουν ψηφιακές υπογραφές και εξασφαλίζουν ασφάλεια. Ευχαριστώ. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Δίνω το λόγο ξανά στον εισηγητή, τον Γιάκομπ Φον Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για καταληκτικές παρατηρήσεις το φάκελο αυτό, όμως οπωσδήποτε θα ήθελα εδώ στο κλείσιμο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πάρα πολύ ευχάριστη εργασία που επιτελέσαμε μαζί. Δεν ήταν μόνο το κλίμα πολύ καλό, αλλά ε, έγιναν και συζητήσεις ενδιαφέρουσες ε, με πολλές προκλήσεις και την επόμενη εβδομάδα είμαι βέβαιος ότι θα παρουσιάσουμε καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες που θα βρουν σύμφωνους όλους. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεργασία. Και εγώ τους ευχαριστώ όλους. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 26 Απριλίου όπως είχε προβλεφθεί και θα πάει στην Ολομέλεια στην δεύτερη σύνοδο του Μαΐου. Και προχωρούμε στο σημείο 7, διεθνή λογιστικά πρότυπα. Δεν θα σας δώσω εγώ εξηγήσεις αφού έχουμε τον ειδικό, τον εισηγητή μας και του δίνω αμέσως το λόγο. Ο Θείοντορ Στόλογιαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά θα ξεκινήσω λέγοντας είμαι ευτυχής που μπορώ να σας παρουσιάσω την έκθεση για την οποία έλαβα ιδέες, προτάσεις από όλους τους σκιοδεσιητές και από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου που υπέβαλαν τις θέσεις τους. Επίσης αξιοποιήσαμε πολλά σεμινάρια, πολλές ακροάσεις, καθώς επίσης και την πανεπίσημη ομάδα εργασίας για τα διεθνή ε, πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς με τη συμμετοχή μελών από όλες τις πολιτικές ομάδες. Όλες τις τροπολογίες που ε, ε, έλαβα ήταν υψηλού επίπεδου. Καταλήξαμε σε 16 συμβιβαστικέ, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο 40 τροπολογίες συναδέλφων και έχουν ήδη γίνει συζητήσεις επί αυτών των συμβιβαστικών ε, τροπολογιών και θα έλεγα ότι μάλλον συμφωνούμε ε, στις περισσότερες από αυτές, για τις περισσότερες από αυτές. Επίσης λάβαμε μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Και θα αναφερθώ στα κυριότερα ζητήματα επί των οποίων προσπαθούσαμε να συμφωνήσουμε. Πρώτα απ' όλα, μία ε, εξπεξήγηση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος. του δημοσίου αγαθού μας, συγχωρείτε. Που συνδέεται με τη σταθερότητα, με την ανάπτυξη. Και αυτή η συζήτηση οδήγησε στη συμβιβαστική τροπολογία Β. Στην τροπολογία C τα ζητήματα της ορθής ε, εκτίμησης και της έννοιας της σύνεσης, η οποία την είχαν διαφορετικών ερμηνεών ανάμεσα στην ICB ε, που καθορίζει ε, αυτά τα πρότυπα, ενώ εμεί έχουμε μια διαφορετική ερμηνεία που προέρχεται από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το τι, τι, τι, τι σημαίνει ε, σύνεση στον δικό τομέα. Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομική αναφοράς επανέρχονται, επαναλαμβάνουν ε, την έννοια της ε, σύνεσης και γι' αυτό στην συμβιβαστική τροπολογία C ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με την ICB για να ε, καταλήξουμε σε έναν καλύτερο ορισμό της σύνεσης. Επίσης, Έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση αντικτύπου. με τη συμμετοχή της συμβουλευτική ομάδας για τα θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς στην ΕΦΡΑΚ ακόμα δεν έχουμε ε, καταλήξει αλλά θα, θα, αναμείνουμε και αυτήν την ε, αξιολόγηση αντικτύπου. Επίσης, στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού γίνεται μια αναφορά στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για τους, διεθνή, ε, συγγνώμη, τους δημόσιους φορείς. Εδώ σημειώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας ειδικό οργανισμός για να καταλήξει σε τέτοια πρότυπα, σε IFRS, σε ε, διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για τον δημόσιο τομέα, τομέα των δημοσίων επιχειρήσεων. Ε, και πρόσφατα διάβασα μια έκθεση, ένα άρθρο για το θέμα αυτό και με έκπληξη διαπίστωσα ότι πολλά παραμένουν ακόμα που πρέπει να γίνουν σε πολλές χώρες. Για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές αναφορές στον ε, τομέα των, των ε, δημοσίων, ε, δημόσιας λογιστικής. Ακόμα μερικοί χρησιμοποιούν χρηματορροές και όχι μεταβατικούς λογαριασμούς. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα ζητήματα ε, θα μπορούσε κανείς να εμπνευστεί από τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για να τα επιλύσει. Συζητήθηκε επίσης πολύ συχνά το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και καταλήξαμε για, ε, από αυτή τη συζήτηση στην ε, συμβαστική τροπολογία H. Γνωρίζουμε όλη τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην τους δημιουργήσουμε ένα υπερβολικό άχθος ζητώντας τους να εφαρμόσουν διεθνή πρότυπα εναρμονισμένα μεταξύ όλων των κρατών μελών τα οποία να εφαρμόζονται με τρόπο ομοιόμορφο σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους. Όταν μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει την Κεφαλαϊκή Ένωση τότε είχε προταθεί να ξεκινήσει μια συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ICB για να καταλήξουμε σε ένα σύστημα διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, το οποίο θα ήταν κατάλληλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι όλες όμως, μόνο εκείνες που σκοπεύουν να εισαχθούν σε κάποιο τύπου ε, χρηματαγορά, όχι το χρηματιστήριο, αλλά σε κάποιο παρόμοιο είδους ε, αγορά. Στη συμβαστική τροπολογία ξεκαθαρίζουμε ότι ένα τέτοιο είδους, μια τέτοιου είδους συνεργασία με την διάθεση την Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεργαστεί με την ICD για να το, για να το επιτελέσει αυτό το έργο, να συνεργαστεί να το κάνει αυτό, Όπω σα είπα ήταν μια ιδέα η οποία προέρχεται από την ιδέα της Ένωσης των Κεφαλαγορών. Τη σημειώνουμε λοιπόν αυτή την πρόθεση της Επιτροπής να το πράξει, αλλά λέμε ότι θα πρέπει οποιαδήποτε ρύθμιση, ε, οποιοδήποτε διεθνές πρότυπο, χρημα... ε, μάλλον, πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς προταθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει σε εθελούσια βάση οι χώρες, τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θέλουν να το υιοθετήσουν ή αν προτιμούν να ακολουθήσουν το δικό τους εθνικό σύστημα. Σε εθελούσια βάση και όχι με νομικά δεσμευτικό τρόπο. Να μπορούν να επιλέξει λοιπόν κάθε κράτο μέλο, εάν επιθυμεί το δικό τη σύστημα ή το σύστημα που από κοινού θα προτείνει η αν προτιμουν να ακολουθησουν το δικο τους εθνικο συστημα σε εθελουσια βαση και οχι με νομικα δεσμευτικο τροπο να μπορουν να επιλεξει λοιπον καθε κρατος μελος εαν επιθυμει το δικο του συστημα η το συστημα που απο κοινου θα προτεινει η κομισιον με την ICB. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο ε, αυτή τη συνεργασία. Υπάρχουν επίση πολλέ άλλε τροπολογίε. για το μέλλον οργανισμών όπως το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων γιατί αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει ε, τακτικά να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διακυβέρνηση του συστήματος αυτού, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, βάση περιπτώσει, και έχουν υπάρξει και κάποιες προτάσεις να μεταβληθεί ε, αυτός ο οργανισμός, να ε, να γίνει κάποια στιγμή ένας διεθνή οργανισμός και νομίζουμε ότι βρίσκουμε μια λύση για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Τώρα, όσον αφορά την ΕΦΡΑΚ, που είναι μια ε, ιδιωτική μη κερδοσκοπική οργάνωση, το Ευρωπαϊκό Συμβουλιο... Ε, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για τα θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς, η ΕΦΡΑΚ λοιπόν, ζητείται ή συζητείται η πιθανότητα να μεταμορφωθεί σε κάποια ευρωπαϊκή υπηρεσία, σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόμοια με την ΕΦΣΑ. Ε, με, κάποια παρόμοια μεθοδολογία. Αναφέρεται λοιπόν αυτό στην έκθεσή μου, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο η ΕΦΡΑΚ κάποια στιγμή να γίνει μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκαθαρίζει ότι σε αυτή τη διαδικασία που ακολουθείται για την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων ε, χρηματοοικονομικής αναφοράς θέλουμε να ε, συνεχίσουμε να συμμετέχουμε και να ενημερωνόμαστε και να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Και θα κλείσω λέγοντας ε, κάτι που συνέβη πριν λίγες μέρες. Δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση της να παραταθεί η χρηματοδότηση της ΕΦΡΑΚ, της συμβουλευτικής ομάδας, και αυτό γιατί όταν είχε αρχικά εγκριθεί ο προπολογισμό ε, με βάση τον οποίο χρηματοδοτείται η ΕΦΡΑΚ, μάλλον ο προπολογισμό με βάση τον οποίο χρηματοδοτείται και η ICB και η ΕΦΡΑΚ και η PIOB, για την συμβουλευτική ομάδα ο χρηματοδότηση έλεγε το 2016. Έλεγε το 2016. Γιατί ο, το πεδίο, η εντολή της ΕΦΡΑΓ ήταν να φροντίσει ε, για την εφαρμογή της ε, έκθεσης ε, και έχουμε και μια ετήσια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της ΕΦΡΑΚ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαρίστω να ακούσω τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, Θεόντορ. Πρώτα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ε, η σκιώδη και η κυρία Περβάος Πέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή μας τον κύριο Στόλογιαν. Γιατί χάρη στην ομάδα εργασίας ε, μπόρεσε να συμπεριλάβει τα σχόλια όλων των συναδέλφων και να τους ακούσει και μάλιστα να τα καλύψει μετά συμβαστικές τροπολογίες που αντανακλούν όλα αυτά τα σχόλια. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σημαντικά θέματα συνεχίζοντας αυτά που είπε ο εισηγητής. Ο εισηγητής μίλησε για κάποιες τροπολογίες, Αιτ Καμάλ και άλλων, που αναφέρονται στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την αληθή και δίκαιη άποψη. Το είπε ο εισηγητής και εδώ θα πρέπει να εξακριβώσω δύο-τρία στοιχεία, να τα ελέγξω, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και στα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σταθώ τώρα σε τέσσερα άλλα σημεία. Καταρχήν, ε, στην έκθεση επιμείναμε να ληφθούν υπόψη κάποιες πτυχές της έκθεσης Μέιστατ. Και επίσης, ε, μια ευρωπαϊκή διάσταση των ε, λογιστικών προτύπων που αναλαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και τους γενικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Και οι συμβαστικές τροπολογίες που συμφωνήσαμε με τον εισηγητή μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερος. Επίσης, ε, αναφέρεται εδώ εν παρόδο μια συζήτηση που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Ε, ο, το ένατο διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς. E ΕΦΡΕΣ 9. Θα δούμε τι θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Πάντως, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές ανησυχίες που αναφέρονται σταδιακά τόσο για τις ε, συνθήκες εφαρμογής ε, του προτύπου 9 στις, ασφάλεις, στις ασφαλίσεις, αλλά και πώς θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις επενδύσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή που δέχτηκε κάποιες τροπολογίες μας. Γιατί, όπω είπαμε, μέχρι στιγμή το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν έχει εκπονήσει μελέτε επιπτώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε σωστές συνθήκες για να προχωρήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί ο εισηγητής μας λέει ότι το θέμα ξαναβγήκε στο φως μετά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, κεφαλαί... την Ένωση Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ε, εδώ και χρόνια κάνει προσπάθεια να πιέσει και να επιβάλλει κάποιες προτάσεις του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμάμαι τον αγώνα που είχαμε κάνει με τον Αλεξάνδρ Άτβαθ, το θυμάστε, ήδη από το 2008, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στη θέση του Συμβουλίου. Δυστυχώ εκτός μικροφώνου το σχόλιο του κυρίου Φέρμπερ. Ναι, αυτό είπα ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. και δεν θέλουμε το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων να εκπονήσει λογιστικά πρότυπα που να τα εφαρμόζει στι μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ και χρόνια το προσπαθεί και θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Ε. Και τώρα θα καταφέραμε να καταλήξουμε συμβαστική τροπολογία με τον εισηγητή που περιγράφει την κατάσταση αντικειμενικά και που κρούει το κόδωνα του κινδύνου για μια ε, δεχόμενη λανθασμένη κατεύθυνση που θα αντιτασσόταν στα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Επίσης, ε, ο εισηγητής είχε την καλοσύνη να συμπεριλάβει και την πρόπτικη της έκθεσης ε, Μάιστα, ώστε η ΕΦΡΑΓ να γίνει μακροπρόθεσμα ένας δημόσιος οργανισμός. Ερωτώ όμως πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμη τα πράγματα με τη συμβαστική τροπολογία Δέλτα. Εκεί που αναφέρεται υπό ποιου όρου θα πρέπει να χρηματοδοτείται η ΕΦΡΑΓ, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για τα θέματα χρηματοοικονομικών αναφορών. Γιατί φαίνεται. Α, συγγνώμη, έκανα λάθο στο... στο γράμμα. Είναι η συμβαστική τροπολογία H, ήτα. Το θέμα είναι ε, να προγραμματίζει ελεύθερα τις εργασίες της η Έχω την αίσθηση όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις των εργασιών της ΕΦΡΑΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν εμπλακεί και στον τρόπο που ε, εκτελεί τις ε, εργασίες της ΕΦΡΑΚ, αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Πρόκειται για τη συμβαστική τροπολογία ενή. Εντάξει, να ζητούμε τη έκθεση από την ΕΦΡΑΚ. Αν όμω δεν έχουμε τα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντλήσουμε συνέπειε από την αξιολόγηση αυτή τη ετήσια έκθεση, τότε θα στερηθούμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο άσκησης επιρροής στην ΕΦΡΑΚ. Και η αιτήσια συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΦΡΑΚ θα πρέπει να συνδέεται με την ετήσια έκθεση. Εκεί θα πρέπει να είμαστε στους πιο κατηγορηματικοί στην συμβαστική τροπολογία νη. Θα υποβάλουμε μια διευκρινιστική πρόταση. Πάντως, κατά του λοιπού, η έκθεση είναι τέλεια. Ευχαριστώ και περνάμε στην ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Έχω την τιμή να, δώσω, να δίνω το λόγο στον Σαΐτ Καμέλ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή, αλλά και τους και οδησηγητές των πολιτικών ομάδων. Μερικές φορές σε κάποια θέματα διαρωτόμαστε αν θα καταλήξουμε ποτέ συμφωνία. Και σε άλλες εκθέσεις όπως αυτή, ήδη από την αρχή έχουμε μεγάλο βαθμό συνένεσης. Και ε, βουλευτές από όλες τις πολιτικές παρατάξεις προβληματίζονται για το θέμα αυτό. Και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία η εικόνα ήταν ομόφωνη σε ό,τι αφορά το χρηματοδότηση της ΕΦΡΑΚ και του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και δεν θα πρέπει να επιτρέπονται υπερτιμήσεις ε, των ε, δαπανών και υποτιμήσεις των εσόδων. Επίσης, θα πρέπει να θεωρηθούν υπόλογοι και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΦΡΑΚ. Και καλό θα ήταν να στήσουμε αυτή την ομάδα εργασία ε, για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικών αναφορών και να είμαστε πολύ αυστηροί στη διαδικασία αυτή. Τώρα έχουμε μια σωστή ισορροπία με την έκθεση, με πολλές τροπολογίες και ε, γενικές συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ ε, θέλω να εξετάζουμε τι λέει ακριβώς ο κανονισμός για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς ε, και να λάβουμε υπόψη την νομολογία του ΔΕΚ, την οδηγία για την κεφαλαϊκή επάρκεια και να το προσέξουμε αυτό στον κανονισμό για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Πάντως, τα λαμβάνει αυτή η υπόψη εισηγητής. Τώρα, διευκρίνηση για το τι συμβαίνει true and fair, δίκαιο και αληθινό, ώστε να έχουμε πραγματικά περιεκτικά κριτήρια έγκρισης. Πάντως, οι συμβαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε μας επιτρέπουν να υλοποιούμε το στόχο μας. Είμαι υπέρ της διατύπωση που εθετήσαμε στις συμβαστικές τροπολογίες και της κατεύθυνση που έλαβαν οι συζητήσει των σκιωδών εισηγητών. Βέβαια, δεν μπόρεσα να εξετάσω διεξοδικά τις τελευταίες τροπολογίες και δεν συμφωνώ εννοείται με όλες τις λεπτομέρειες. Μερικά θέματα ακόμη με προβληματίζουν. Πάντως δεν υπάρχουν πολλές διαφωνίες και θα φανεί αυτό και στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ευχαριστώ, Σαγέντ. Εκπρόσωπο των φιλελευθέρων δεν βλέπω από τους και ηγητές, οπότε εκ μέρους συγκούε, Γκουε, ο Φάμπιο Ντεμάζη. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά. Και εγώ προσυπογράφω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι είχαμε καλή και επικοδομητική ατμόσφαιρα εργασίας εξετάσαμε την πρόταση που υπευλήθη πρόσφατα από τον ο Καμάλα για το True and Fair, τις γραμμές του δικαστηρίου και βεβαίως ε, χρησιμοποιήσαμε ένα στρατό δικηγόρων ε, αν και ε, είναι... και αποφύγαμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε, στρατόδικηγόρων γιατί βασιστήκαμε στη γνώμη του που είναι εμπεριστατωμένη. Εμείς έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις. Θα πρέπει να γίνει δημόσια ω οργανισμός η ΕΦΡΑΓ. Επίση ε, θα πρέπει να έχουμε ε, διεθνεί, διεθνείς δημόσιους οργανισμούς ε, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και από σειρά εμπλεκομένων όπως εκπροσώπους ε, ε, επιχειρήσεων, κοινωνίας των πολιτών. άλλα θέματα θα πρέπει να τα χειριστεί η ειδική έκθεση και, και, και το, βεβαίως για το πρότυπο 9 και το ρόλο του, των διεθνών προτύπων στη φοροδιαφυγή υποβολή εκθέσεων αναχώρα επίσης είναι σημαντικό και το ε, πρότυπο 9 εδώ κάποιοι έχουν τη γνώμη ότι ίσως δεν είναι ο σωστός τόπος και χρόνος για να το εξετάσουμε αυτό το θέμα και να το λύσουμε. Θα διατηρήσουμε τις δύο σχετικές τροπολογίες μας γιατί πρόκειται για θέμα αρχής χωρίς όμως αυτό να υπονομεύει την σύμφωνη γνώμη που θα εκφράσουμε για το ψήφισμα. Επίσης μπορούμε να έχουμε βελτιώσεις ακόμα επί δύο συμβιβαστικών τροπολογιών η ΕΝ που λέει τώρα καλεί την Κομισιόν να αξιολογήσει την δυνατότητα και πιθανότητα να δημιουργηθεί δημόσιος οργανισμός ούτως ώστε μακροπρόθεσμα να αντικατασταθεί η ΕΦΡΑΓ η ομάδα Άλντε είπε ότι θα μιλούσε για μετασχηματισμό και όχι αντικατάσταση της ΕΦΡΑΓ. Αυτό είναι εντάξει, δεν μας πειράζει. Όμως αντί να πούμε να, αξιολογήσει, να, αξιοποιήσει, αξιολογήσει τη δυνατότητα δημιουργίας δημοσίου οργανισμού, ίσως μπορούμε να πούμε καλή την Κομισιόν να αναπτύξει μηχανισμούς μετασχηματισμού της ΕΦΡΑΓ μέσω πρόθεσμα ώστε να γίνει δημόσιος οργανισμός, αλλά αυτό μπορεί να το εξετάσει ο εισηγητής μάλλον και θα βρούμε συμβαστική λύση. Για τη συμβαστική H θα θέλαμε να διατηρηθεί η τροπολογία 67 του Σφεν Γκίγκολτ που λέει ότι είναι πεπισμένος ότι δεν συνδικάτα, οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, τα Υπουργεία Οικονομικών θα πρέπει να ε, εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Αν δεν είναι δυνατό, εναλλακτικά προτείνουμε να ε, έχουμε μια σειρά εκπροσώπων ε, ε, συμφερόντων στην τροπολογία 35 και να πάει στην συμβιβαστική W αν δεν μπορεί η αρχική τροπολογία Giggle να διατηρηθεί στη συμβιβαστική H. Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές παρατηρήσεις, τα άλλα είναι εντάξει. Εντάξει, ο Σβέν Γκίγκολτ. Να ευχαριστήσω και εγώ θερμά τον κύριο Στόλογεν και όλη την ομάδα. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία και γενικά θέλω να ε, πω ότι μετά τους συναδέλφους ε, Περέζ και Καμάλ οι τροπολογίες κινήθηκαν προς παρόμοια κατεύθυνση. Δεν είχαμε θεμελιώδεις διαφορές. Οπότε θα ήθελα αυτή τη σύντομη συζήτηση να την αξιοποιήσω αναφερόμενος στις τροπολογίες της κυρίας Κάπελ κυρίως από το Αυστριακό κόμμα, Λαϊκό Κόμμα, γιατί μου κάναν κατάπληξη ορισμένες. Δηλαδή δεν ταιριάζουν, είναι εκτός τόπου. Ε, η κυρία Κάπελ ε, συνολικά λέει ότι θα πρέπει τα πρότυπα να επεκταθούν ακόμη περισσότερο και μάλιστα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κυβερνητικούς οργανισμούς. Ε, θέλει να εφαρμόζονται παντού τα πρότυπα, τα πρότυπα αυτά και αυτό εκπλήσει γιατί κατά τα άλλα στην Αυστρία η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνεται ως αντιδημοκρατική, ενώ ε, το Διεθνές Συμβούλιο, όπου η δημοκρατία και οι εκλογές είναι ε, ξένη λέξη, θα πρέπει να επιβάλλει πρότυπα σε όλη την Ευρώπη. Ε, Ω ομάδα εργασία που ασχοληθήκαμε πολύ για το θέμα, συζητούσαμε πάντα αν η αρχή του true and fair, δηλαδή τη ορθότητα και τη αμερόληπτη απεικόνηση, ε, καλύπτεται από τα διεθνή πρότυπα αυτά. όλες Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Ε, υπάρχουν κάποιες παραδόσεις σε σχέση με τους απολογισμούς που δεν, δεν είναι ταυτόσιμοι με τα πρότυπα εδώ. Άρα λοιπόν ε, τα κέρδη ε, θα, θα πρέπει ε, να δικαιολογούνται και να αναλύονται. Αυτό αυτή η ανάγκη, αυτή η αρχή δεν καλύπτεται. Ε, και ορισμένα πράγματα ε, ε, τα δέχεται χωρίς καμία κριτική. Πώς θα εξηγήσετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον τρόπο δήλωσης των εσόδων και κερδών ε, δεν θα μπορούσαν να το καταλάβουν ε, και βλέπω και αντίφαση στον προσανατολισμό που έχετε στην Αυστρία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί ε, τους λέτε πολλά θετικά ενώ εδώ παίρνετε θέση υπέρ αρχών που δυστυχώς ε, δεν καλύπτουν τις πρακτικές ανάγκες. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και δημόσια όταν υποβάλετε τροπολογίες που δεν ταιριάζουν με την κατά τα άλλα ρητορική του κόμματός σας. Ευχαριστώ. Από την EFTD δεν έχουμε ε, σκιώδη. Περνάμε στην Μπάρμπαρα Κάπελ από το ΙΕΝΕΦ. E ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι που μου δώσατε το λόγο για να απαντήσω. Ε, ε, ευχαριστώ τον κύριο Γκίγκολτ που ασχολήθηκε με τις τροπολογίες του κόμματός μας που είναι ισχυρότερη με το 33%. Ε, βεβαίως και δίνουμε προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και εγώ ασχολούμαι ιδιαίτερα με το θέμα και χαίρομαι που ασχοληθήκατε κι εσείς. Θα ήθελα να πω ότι όταν μιλάμε για διεθνή λογιστικά πρότυπα ε, θα πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια προοπτική. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε ε, πρότυπα ε, αποδεκτά όπως είναι μέχρι τώρα από 116 χώρες. Οι μεγάλες αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις ανάλογα με την κεφαλαιακή τους ε, κάλυψη ε, θα πρέπει να μπορούν να κινούνται και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτά είναι γενικότερες αρχές απόλυτα αποδεκτές και αντικατοπτριζόμενες και στο πρόγραμμα του κόμματος εαυτός Εγώ συμμετείχα στην κατάρτιση του προγράμματος και το γνωρίζω. Κατά τα άλλα είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αξιολογήσεις και εν προκειμένου η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική. Ε, ο σχετικός κανονισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα πλαίσια της ρύθμισης ε, και στις δημοσιονομικές υπηρεσίες. Ε, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ΕΚΑ ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή εργασία του. Οι 16, 16 τροπολογίες είναι ε, βελτιωτικές και πιστεύω ότι είναι θετική αυτή η ε, έκθεση ε, πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι έγινε δυνατόν να ε, αντιμετωπιστεί η μεγάλη συνθετότητα και περιπλοκότητα των ε, χρηματοοικονομικών αγορών, ε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου έχουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτήν την προαιρετική χρήση των προτύπων. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό το στοιχείο του προαιρετικού είναι πολύ σημαντικό στην τροπολογία. Ε, η συνοχή, η συνέπεια, ε, πιστεύω ότι ε, ελήφθησαν υπόψη επαρκέστατα. Ο στόχος είναι το Διεθνές Συμβούλιο να εγκρίνει και να ε, ε, διασφαλίσει διεθνή πρότυπα τα οποία θα μπορούν ε, παγκόσμια να γίνονται δεκτά. Επίσης θα πρέπει να, είναι και ισο... να υπάρχει ισοτιμία και με τα πρότυπα άλλων χωρών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν τον Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων τους των Ηνωμένων Πολιτειών και πρέπει αυτά να λυθούν υπόψη στην ε, συμβιβαστική λύση, προπολογία ε, Β επίσης ε, όλα αυτά ρυθμίζονται καλά, όπως και στην συμβιβαστική N που η μεταρρύθμιση ε, μας βρίσκει σύμφωνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο. Οπότε να ξαναδώσω το λόγο στον Θεότρο Στόλογεν για τα τελικά του σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα στα σχόλια των συναδέλφων και θα σταθώ σε λίγα θέματα για τα οποία έχουμε μερικές διαφωνίες. Η κυρία Μπερές είπε σαφώς ότι θα πρέπει να έχουμε και, και μια μαγκούρα ε, στους φορείς που χρηματοδοτούμε για να επηρεάσουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αναφέρθηκε και απευθεία στην ΕΦΡΑΓ, ώστε να, και είπε να συνδέσουμε τη χρηματοδότησή μας με την ετήσια έκθεση της ε, μεταρρύθμισης που εφαρμόζει η ΕΦΡΑΓ, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Κατά τη γνώμη μου, ε, η ΕΦΡΑΓ έχει πολλούς κορυφαίους εμπειρογνώμονες Και εμείς θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη θέση για τη χρηματοδότηση. Μάλιστα, αν δεν έχουμε σαφή θέση για τη χρηματοδότηση, άκουσα από την ΕΦΡΑΚ ότι μερικοί εμπειρογνώμονες θα ζητήσουν αλλού δουλειά. Βέβαια αυτό είναι θέμα της ΕΦΡΑΚ περισσότερο, να τους κρατήσει. Πάντως κυρία Μπερές, ήδη έχουμε λάβει το σχέδιο κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της ΕΦΡΑΚ θα πρότεινα να υπερψηφίσετε τη συμβαστική τροπολογία και όταν, λάβουμε την, και όταν έχουμε την έκθεση για την παράταση της χρηματοδότησης ΕΦΡΑΓ για την τριετία 2017-2020 να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Επευκαιρία της έκθεσης για την ΕΦΡΑΚ και την παράταση της χρηματοδότησης. Τη περίοδου χρηματοδότηση. Αυτή είναι η πρότασή μου. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμφωνώ απόλυτα με του συναδέλφου. Και να σας εξηγήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε αυτό το θέμα στο ζήτημα της ε, ε, Ένωσης Κεφαλαγορών. Γιατί όταν μιλούμε για Ένωση Κεφαλαγορών, Μιλούμε και για διαφορετικές οργανωμένες αγορές, όπου μερικέ μικρομεσαίες επιχειρήσει θα είναι εισηγμένε. Υπάρχουν άλλου είδου ε, ε, οργανωμένες αγορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Λόρδο Χίλε και, θα συζη... Ε, που εξέταζαν την Ένωση Αγορών σκέφτηκαν να υιοθετήσουν παρόμοια αντίληψη και για, τις, για τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως εμείς εμένουμε στη δική μας θέση ότι οποιαδήποτε αποτέλεσμα αυτών των εργασιών ισχύει μόνο προαιρετικά ε, οικειοθελώς ε, και να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι αυτό το σχέδιο των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, αν προβλέπονται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι υποχρεωτική εφαρμογή. Επίσης θα προσπαθήσω με τον βοηθό μου να συμπεριλάβω και κάποιες προτάσεις που την τελευταία στιγμή μας έστειλαν οι φίλοι ελεύθεροι. Μερικά σχολεία τους είναι εύστοχα και μπορούμε να τα καλύψουμε στις συμβαστικές μας τροπολογίες. Μια και δεν αλλάζουν την ουσία τους, αλλά διευκρινίζουν κάποια επιμέρους σημεία. Γι' αυτό θα συμπεριλάβω στις συμβαστικές μου τροπολογίες κάποιες ε, αλλαγές τελευταία στιγμή που πρότειναν οι φιλελεύθεροι. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Και ευχαριστώ και τους και ηγετές για το έργο τους. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στην ψηφοφορία, γιατί έχει προβλεφθεί για τις 25 και 26 Απριλίου την επόμενη μας συνεδρίαση. Θα δούμε αν και κατά πόσο θα στηριχθούν και θα υπερψηφιστούν οι συμβαστικές τους τροπολογίες. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 8 της ημερήσης διάταξης, τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ετήσια έκθεση για το 2014. Δεν βλέπω όμως τον εισηγητή μας, τον κύριο Τρεμόζα Ιμπαλσέλς. Έχει κανείς από τους φιλελεύθερους ε, καμιά ιδέα που βρίσκεται ο Ραμόν αυτή τη στιγμή ή κάποιος υπάρχει που μπορεί να τον αντικαταστήσει μήπως για το σημείο 8. Ξέρω ότι <laughs> είμαστε ένα λεπτό νωρίτερα, μα άμα έχετε Γερμανό πρόεδρο αυτά παθαίνετε. Ε, λειτουργούμε με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού τι να κάνω τώρα, να ανοίξω τη συζήτηση χωρίς ε, να έχουμε ακούσει την ενημέρωση και ερήμην του εισηγητού, του συντάκτη γνωμοδότησης. Προσπαθούμε, τον ψάχνουμε στο γραφείο του, δεν ξέρω που ακριβώς είναι. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το γραφείο του. Τι να κάνουμε, πεντάλεπτο διάλειμμα, δίλεπτο. Α, καταφθάνει. Άρα ένα λεπτό διάλειμμα είναι αρκετό. Γιατί τον περιμένουμε να στη στιγμή τώρα μόνο. But I was a little bit in advance, two minutes before five. Uh, we've been ready Προλάβαμε και ολοκληρώσαμε τα προηγούμενα θέματα δύο-τρία λεπτά νωρίτερα. Πάντω, ευχαριστούμε που ήρθατε εσεί καιρό και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 8 τη ημερήσια διάταξη, τον έλεγχο τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη έκθεση για το 2014. Με χαρά και τιμή δίνω το λόγο στον συντάκτη της γνωμοδότησής μας, τον κύριο Ραμόν Τε... Τρεμόσα Ιμπαλτζέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ νιώθω μεγάλη τιμή που είστε εσείς πρόεδρος σήμερα. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε την περασμένη Τετάρτη στο Στρασβούργο την πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών επί του κειμένου που σας είχα στείλει την περασμένη εβδομάδα. Ε, έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το ECR με ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δεν μπορώ βέβαια να σας υποσχεθώ ότι θα τις κάνω όλες δεκτές, αλλά σίγουρα τις περισσότερες. Θα προσπαθήσω να τις καλύψω γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες DH, I και J. Ευχαριστώ λοιπόν την ομάδα μεταρρυθμιστών και συντηρητικών και την Κέι που μου έστειλε και γραπτός ένα ε, ηλεκτρονικό μήνυμα με τις προτάσεις, αλλά άλλο κανεί δεν μου στείλε προτάσεις. Βέβαια, ήταν και μικρό το διάστημα. Αύριο θα ξανασυνεδριάσουμε με τους σκιώδεις ηγητές και πιστεύω ότι θα πραγματοποιήσουμε σημαντική πρόοδο, γιατί όλοι οι σκιώδεις είχαν στο μεταξύ το χρόνο να θέσουν τα ζητήματα στις πολιτικές τους ομάδες και να καταλήξουν σε πολλά σημεία συμφωνίας. Έχουμε ένα πρόβλημα από την άποψη ότι η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου δεν είναι όπως θα έπρεπε. Έχουμε εκατοντάδες έως και χιλιάδες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, διαδικασίες επιπαραβάση που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία τετραετία. Περίπου 4.000 τέτοιες υποθέσεις έχουμε και χίλιες περίπου το χρόνο. Έχουμε πρόβλημα και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, καταλαβα... δεν καταφέρει να πει στα κράτη-μέλη, να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν πλήρως την εσωτερική τους ένωμη τάξη και να εφαρμόσουν το ενωσιακό δίκαιο, τότε χάνουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αξιοπιστία μας. Και ίσως ε, είναι και ένας από τους λόγους της έξαρσης ε, του, ευρωσκεπτικισ... ευρωσκεπτικισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πρόβλημα το αισθανιζόμαστε όλοι, το έχουμε αναγνωρίσει όλοι και έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις. Μία ήταν να συστήσουμε μία υποεπιτροπή για να εξετάσουμε αυτά τα επιμέρους ε, θέματα, δηλαδή πώς ε, μεταφέρεται το ενωσιακό δίκαιο στα κράτη-μέλη και να, κάνουμε, να εξασφαλίσουμε μια παρακολούθηση του θέματος. Αυτή η υποεπιτροπή θα μπορούσε να είναι υπό την αιγύδα της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ΑΦΚΟ ή Γιούρι είναι προσυζήτηση αυτό. Οι φιλελεύθεροι επίσης προτείνουν να συμπεριλάβουμε στη συζήτηση και βασικά τραπεζικά ιδρύματα για να μας βοηθήσουν. Δεν ξέρω, Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, ε, Τραπεζών, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν ξέρω ποιος. Πάντως το θέμα είναι να υπάρχει μια λογοδοσία για το πώς εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο στα κράτη-μέλη. Μία πρόταση κάνω. Ας ε, συζητήσουμε τι τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να μας βοηθήσουν ή τι τραπεζικά ιδρύματα. Περιμένω τις απαντήσεις σας και τις αντιδράσεις σας και τα σχόλιά σας. Μέχρι αύριο, που θα είναι η δεύτερη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών, ελπίζω να τα βρούμε, να συνεννοηθούμε και να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα όπως προβλέπεται στο πρόγραμμά μας. Θα μας πει και η γραμματεία αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Πάντως πιστεύω ότι αν καταλήξουμε γρήγορα σε συνένεση θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν. Θα ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις συζητητές. Κύριος από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την δουλειά του έως τώρα. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί να συζητήσουμε περισσότερο και με τον συντονιστή μας για να βρούμε μια συμφωνία. Η ΕΛΚ έχει ε, υποβάλει ε, πολλές τροπολογίες, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, αναφερόμαστε στην οικονομική κρίση, αναφερόμαστε στο δημόσιο χρέος. Αύριο θα γίνει μια πολύ σημαντική συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και νομίζω ότι σε αυτήν θα καταφέρουμε να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε σχεδόν σε όλα. αλλά επίσης αύριο αναμένω να ακούσω και τις δικές σας α, ε, απόψεις για το ποιες θα είναι, ποια θα είναι η θέση μας στο, ε, στη διαπραγμάτευση. Ο κύριος Φρουντσούλητσα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω όλους εδώ για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, συγχαίρω τον εισηγητή και όλους τους άλλους σκιώδεις. Όσον αφορά τις τροπολογίες και τις συμβιβαστικές τροπολογίες, πρέπει να σας πω ότι παραμένουν ακόμα διαφορές. Ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, που, συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες θα θέλαμε να έρθουν πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Αύριο θα γίνει το απόγευμα μια συνάντηση των σκιωδών, αλλά δυστυχώς εγώ πρέπει να αποχωρήσω γιατί πέμπτη πρωί πρέπει να είμαστε μια πολύ σημαντική πολιτική συνάντηση στο Βουκουρέστι. Θα πρότεινα λοιπόν, εάν γίνεται, να συναντηθούμε μεσημέρι ή το πρωί. Εάν όχι, θα σας στείλω τη θέση μας για τις συμβαστικές τροπολογίες γραπτός μέσω email. Για όλες τις συμβαστικές που έχετε προτείνει. Εγώ θα ήθελα και πάλι να τονίσω τα εξή λέμε ότι η έλλειψη εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου συνέβαλε σε διάφορες από τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι επίσης έχει οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Επίσης αναγνωρίζουμε ότι η βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα αύξανε και την εμπιστοσύνη που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στην Ένωση τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμφωνούν σε ένα πιο ε, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την θέση σε ισχύ και την εφαρμογή των νομοθετημάτων, για να μπορούν και τα κράτη-μέλη να, τα εφαρμόζουν. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουν ότι οι 11 οδηγίες που αφορούν ε, στα θέματα αυτά τα χρηματοοικονομικά και ακόμα δεν έχουν μεταγραφεί από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη θα υλοποιηθούν, θα γίνει αυτό επιγόντως. Ο εισηγητής ε, λέει ότι η μη σωστή εφαρμογή του συμφώνου ε, σταθερότητας ε, οδήγησε στην κρίση του 2008. Αλλά, κανείς δεν, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτή την προσέγγιση λεσεφέρ που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα, το οποίο βέβαια το καταλαβαίνω γιατί τους φιλελεύθερους αυτή η νοοτροπία είναι σημαντική είναι, την υιοθετούν. Ε, το κανονιστικό πλαίσιο είναι σημαντικό και χαίρομαι που αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή διάσταση του συστήματος εγγύησης καταθέσεων, αλλά θα πρέπει να βεβαιώσουμε ότι δεν ε, επιδιώκουμε και αντιφατικούς στόχους με αυτό το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Οι κυρώσεις ε, θα πρέπει να γίνουν περισσότερο αναλογικές και περισσότερο αυστηρές για εκείνα τα κράτη-μέλη, ιδίω εκείνα τα οποία συστηματικά δεν εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, για τα οποία υπάρχουν πολλές διαδικασίες επί παραβάση ανοιχτές. όταν έχουμε ένα νομοθέτημα, ε, ε, μάλλον το όταν αναφερόμαστε σε μια διαδικασία και αναφερόμαστε στην έκθεση για σε κάποιε χώρε που δεν την έχουν εφαρμόσει για σε μια διαδικασία επιβαρεβάση η οποία έχει ξεκινήσει, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να αναφέρουμε ονομαστικά όλε τι χώρε, όχι να λέμε μόνο δύο ή τρει ή τέσσερι από αυτέ, ή να μην αναφερόμαστε σε κανέναν. Θα πρέπει η Κομισιόν να είναι ξεκάθαρη ε, ως προς το ποια κράτη-μέλη δεν ε, σέβονται την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Και πάλι σα ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία μου με τους ε, συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και στα Ιταλικά. Φέρουμε στην πολυγλωσία. Grazie Presidente. Um, uh, I'm, I'm, ah, okay. I'm speaking. Uh, I'm speaking here on. Είμαι εκπροσωπό των Κέι Φούιμπερ που δεν μπόρεσε να έρθει εδώ δυστυχώς. Τι συνάδελφο ε, είχε κάποια σύντομα σχόλια να κάνει και για τι συμβιβαστικέ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρεί τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά ανέφερε που έχουν αποτύχει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις οδηγίες της Ένωσης και πιστεύει ότι στο βαθμό που γίνεται κατονομάζονται και ντροπιάζονται, αυτό είναι καλή προσέγγιση από την Κομισιόν. Σωστό είναι να μπορούμε να κατονομάζουμε τους χειρότερους παραβάτες και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν πότε οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται. Ε, οπότε εδώ δεν συμφωνούμε με τον σκιώδη της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Δεν υποστηρίζει όμως του τομεί της έκθεσης που αναφέρονται σε μελλοντική νομοθεσία ή κείμενα που ακόμη δεν έχουν συμφωνηθεί. Είναι πιο ενοιολογικά ή θεωρητικά ή καθοδηγητικά. Οι συστάσεις αναχώρα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι συστάσεις. Θα ήταν παράξενο να έχουν το, την ίδια ισχύ όπως οι οδηγίες στην έκθεση αυτή. Αυτές οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές και θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι είναι. Και αυτό αληθεύει ακόμη περισσότερο αν δούμε και τα διεθνή πρότυπα. Αλλά εκτός από αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετική η ε, έκθεση και περιμένει με ενδιαφέρον την περαιτέρω συνεργασία και με τον εισηγητή και τους άλλους συναδέλφους για να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Μαθ Κάρτιν για την Γκουε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή που προσπάθησε πολύ να διασφαλίσει όσο γίνεται πιο ευρεία πολιτική υποστήριξη της έκθεσης. Εκτιμώ τις προσπάθειες του εισηγητή. Ε, εξήγησα στη συνεδρία των Σκιωδών ότι καμιά φορά η γέφυρα και το... η ε, διαφορά μεταξύ μας είναι πολύ μεγάλη. Αυτό έχει να κάνει με θεμελιώδεις αρχές διαφωνίας σχετικά με το πώς προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά και τη θετική ή μη ε, φύση του ενωσιακού δικαίου και του αντίκτυπου που έχει στις διάφορες χώρες. Εγώ είμαι πεπισμένος και το έχω πει ότι αποφάσεις ε, που αφορούν τις κοινότητες πρέπει να, γίνουν, να λαμβάνονται κοντά στις, κοινότητες, στις μικρές αυτές κοινότητες, ενώ το ενωσιακό δίκαιο το ξεπερνάει αυτό το όριο. Όταν ε, βλέπουμε επίσης την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου πρέπει να κοιτάμε και τις επιπτώσεις του δικαίου ή των νόμων. Σημείωσα για παράδειγμα και το, ε, ανέφερα και στους κοιόδης, ότι όταν Μιλάμε για τραπεζικό τομέα και νομοθεσία στα χρηματοοικονομικά. Μόνο η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις ε, νομοθετικές απαιτήσεις. Ένα θεμητό ερώτημα είναι αν το ενωσιακό δίκαιο ε, καλύπτει και ταιριάζει σε κάποια κράτη-μέλη περισσότερο από ό,τι ε, άλλα. Καμιά φορά οι νόμοι που εγκρίνονται εδώ και από άλλα θεσμικά όργανα επέδρασαν επιβλαβώς ιδιαίτερα σε περιφερικές χώρες και τις χώρες που ε, μπήκαν σε προγράμματα bailout. Ε, μετά την αρχική συνάντηση προέκυψαν συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχει περιθώριο ευρεία συμφωνίας. Έχουμε παρουσιάσει ορισμένες πολιτικές παρατηρήσεις και ε, έχουν ληφθεί υπόψη αρκετές. Εκεί θα χαρούμε να ψηφίσουμε υπέρ. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω στη συνάντηση των σκιωδών αύριο γιατί πρέπει να γυρίσω στην Ιρλανδία. Αλλά η Γκουέ θα εκπροσωπηθεί ε, από κάποιον συνεργάτη μας ε, και ελπίζω ότι εκεί όπου έχουμε έγκυρα επιχειρήματα θα ληφθούν αυτά υπόψη. Η κατεύθυνση που ακολουθεί η έκθεση αυτή ε, έχει να κάνει με την αποκάλυψη τομέων όπου οι νόμοι δεν εφαρμόστηκαν και δεν θα είχα ε, πρόβλημα να αναφερθούν κάποιες χώρες. Γιατί να το φοβόμαστε αυτό ως θέμα αρχής. Και σίγουρα σε κάποιους τομείς η, ανα, ε, ε, ονομασία, κατονομασία αυτών των χωρών θα μπορούσε να έχει θετικό αποτέλεσμα. Να ξέρουμε που οι εθνικές κυβερνήσεις δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί να αποκαλυφθούν και θεμελιώδη προβλήματα της ίδιας της νομοθεσίας. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνάντηση των σκιωδών αύριο. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους δεν βλέπω κανέναν. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, ο πρόσωπος των ε, προσύνων δεν είναι εδώ, αλλά εν πολύ συμφώνησε με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Προς τον συνάδελφο από τη ρουμανική ομάδα θα πω ότι ε, αύριο μπορώ να βρω χρόνο για μια διμερή συνάντηση. Θα το τσεκάρω για να δούμε πότε. Ευχαρίστως να συναντηθούμε διμερώς και να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε κάπου. Μην φύγετε, περιμένετε. Μην φύγετε όπως έφυγε ο κ. Μαλτουτσέλο για να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν βέβαια πολύ πιο εύκολο για όλους μας και για μένα να πούμε εντάξει, ας μην αναφέρουμε κανένα όνομα κράτους μέλους σε αυτή την έκθεση. Αυτό θα ήταν μια εύκολη λύση και θα τελειώναμε σε ένα λεπτό. Είναι και αυτό μια επιλογή. Και βέβαια, αν η πλειοψηφία των βουλευτών σε αυτή την επιτροπή πουν μην το παίξετε αυτό το παιχνίδι του, της κατονομασίας κάποιας χώρας, μην αναφέρετε το, τα ονόματα που είναι στον κακό κατάλογο, γιατί μπορεί κανείς να τα ονομάσει και να τις ε, κάνει να ντραπούν, μπορεί όμως να τις ονομάσει για να τις επενέσει, είναι και ο θετικός κατάλογος. Θα ήταν πιο εύκολο βέβαια να κάνουμε ό,τι κάνουμε συνήθως. Να πούμε ναι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν λαμβάνει υπόψη η ενωσιακή νομοθεσία στα κράτη-μέλη, αλλά ε, να πούμε δύο ωραία λόγια και να συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι από καιρούς καιρό πρέπει να λέμε και κάποιες αλήθειες. Και όχι να λέμε μόνο, να κάνουμε ε, γενικές, ε, να βγάζουμε λόγους, αλλά να αναφέρουμε και κάποιες χώρες που άλλωστε αναφέρονται και στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού βρίσκονται εκεί τα ονόματα, γιατί να μην τα αναφέρουμε και εμείς, γιατί να μην αναφέρουμε ονόματα χωρών. Έχουμε πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες, γιατί θα πρέπει να τις βγάλουμε έξω ε, από την έκθεση. Αύριο το μεσημέρι μάλλον θα γίνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση του Επιτρόπου Βεστάγκεν ε, κατά της Google του Google. Ήμουν ε, ε, εισηγητής στην έκθεση για τον ανταγωνισμό και υπήρχαν κάποιες αποδείξεις ε, ή κάποιες ενδείξεις ότι η Κομισιόν όπως το 2015 θα έκανε μία δήλωση ε, ένστασης κατά της Google σε μια, μια διαδικασία αντιτράστ. Και το ερώτηση, το ερώτημα ήταν έπρεπε να αναφερθεί ρητά το όνομα της Google στην έκθεση ή όχι. Και μετά από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, το θυμάμαι, 600 ε, βουλευτές στην Ολομέλεια ψήφισαν υπέρ του να αναφέρομαι την Google, διότι έχει 90% του μεριδίου αγοράς ως ε, μηχανή έρευνας στις ε, όλες σχεδόν τις χώρες μέλη. Και τώρα έχουμε το ίδιο με το Android. Ε, αύριο το μεσημέρι θα δούμε λοιπόν τι θα πει η Κομισιόν και ε, πώς θα προχωρήσει, θα κάνει δεύτερη δήλωση ένστασης κατά της ε, Google για το Android. Εμείς πριν από τρία χρόνια κάναμε τη δουλειά που έπρεπε γιατί ε, εστιάσαμε σε μια εταιρεία η οποία παραμέριζε τις ευρωπαϊκές. Είμαι υπέρ της αναφοράς στα ονόματα των χωρών που έκαναν καλή δουλειά προκειμένου περί της εφαρμογής του νοσιακού δικαίου και από την άλλη ασκούμε και πιέσεις στις χώρες εκείνες που ακόμα δεν έκαναν αυτά που πρέπει. Η ανα... Αν δεν κάνουμε name and shame θα δημιουργήσουμε περισσότερους κινδύνους εδώ. Βέβαια αυτή είναι μια γνώμη. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Εδώ είμαστε δημοκράτες. Θα δεχτώ εγώ το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας και θα, έτσι θα συνεχίσουμε. Πάντως ε, γι' αυτό ήθελα να γίνει αυτή η συζήτηση και να ακούσω τη γνώμη σας γιατί είναι, θα είναι καλή η συνεισφορά μας νομίζω αν μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν κατάλογο και να βάλουμε μέσα εκεί τις χώρες που κάνουν τη δουλειά όπως έπρεπε και τις χώρες που δεν έχουν κάνει ακόμα τη δουλειά που πρέπει. Λοιπόν, στο Σάντερ Λούνες ναι, την περασμένη εβδομάδα είπαμε ναι στην Κέι Σουίνμπουργκ. Δεν έχει νόημα να αναφέρομαι ενωσιακό δίκαιο που δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει θεσπιστεί, οπότε αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Είχε δίκαιο η Κέι εδώ και άλλες ομάδες συμφώνησαν επίσης. Οπότε αυτό που αναφέρατε θα ληφθεί υπόψη. Και για τον συνάδελφο από την ομάδα Γκουε, αν θέλετε να συναντηθούμε, αύριο το πρωί μπορούμε να βρούμε κάποιο χρόνο. Και αύριο το απόγευμα ελπίζω να είναι σύντομη και όχι μακρά η συνεδρίαση των σκιωδών, ούτως ώστε να ε, διατηρήσουμε και το πρόγραμμα που έχουμε για την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία... η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ θα γίνει στις 26 Απριλίου. και στην ε, Επιτροπή στις 24 Μαΐου και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Ελπίζω λοιπόν μετά τη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών να καταλήξετε σε ε, μεγάλη υποστήριξη του κειμένου του συμβιβαστικού στο οποίο θα καταλήξετε. Έχουμε τελειώσει 6 λεπτά νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Και πρέπει να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη, αν είναι όλοι εδώ. Η Σιλβή ναι, ο Σάντερ ναι, ο Δημήτρη ναι. Έστερ, συμφωνείτε ότι μπορούμε να περιμένουμε λίγο μέχρι τις 5.30 που ήταν και ο χρόνος που είχε προγραμματιστεί. Να ξεκινήσουμε τότε στις 5.30, επομένως 5 λεπτά διάλειμμα παρακαλώ. But don't go away. Αλλά μην φύγετε από την αίθουσα. Eh, eh sono riuscito, ho dovuto un casino. Com'è andata? Dear colleagues, we can start uh, with the vote. Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να περάσουμε στη ψηφοφορία. Όχι, πλάκα κάνω. Θα δοκιμάσουμε. Όχι, όχι. So we have this second exchange of views. Continuing from the last... Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας μετά από την συζήτηση που είχα κάνει στις 7 ε, Απριλίου θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια Λάγκεν Είναι η τρίτη συζήτηση λοιπόν που... Θα κάνουμε μεταξύ έχουμε συζητήσει πολλές φορές μεταξύ μας με διάφορα από τα ενδιαφερόμενα μέρη και εδώ διαπιστώνουμε ότι συγκρούονται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πλειονότητα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το βλέπουν το ζήτημα ως περισσότερο ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους πολίτες, τους καταναλωτές. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αδικία εξαιτίας του ότι τι θα σου συμβεί εξαρτάται από το που, έχει κανείς ε, τις καταθέσεις του, από το ε, ε, που έχει γεννηθεί τελικά, που έχει τα χρήματά του, από αυτό εξαρτάται εάν είναι ασφαλή ή όχι. Αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις με τους συναδέλφους. Όταν πάλι συζητώ με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου αναφέρουν ότι το σημαντικό ζήτημα είναι ότι ακολούθησαν το άρθρο, ε, ε, επέλεξαν το άρθρο 114 της συνθήκης ως την νομική βάση και άρα το ζήτημα είναι περισσότερο ζήτημα οργάνωσης της αγοράς. Και πάλι είναι μεγάλη συζήτηση για το εάν αυτό το άρθρο ήταν το καταλληλότερο. Εν πάση περιπτώσει. Τα κράτη-μέλη θεωρούν περισσότερο ότι το ζήτημα είναι ζήτημα διακυβέρνησης πώς θα ε, εξασφαλιστεί η παρέμβαση του κράτους σε αυτές τις περιπτώσεις. Και φαντάζομαι ότι στο τέλος θα βρεθεί μια συμβαστική λύση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης ανάμεσα σε αυτές τις τρεις προσεγγίσεις. Όπως σας είχα πει, προσπαθούμε να δείξουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε και ποιες είναι, ποια, άλλα θέματα συνδέονται ζητήματα συστημικού χαρακτήρα της Τραπεζικής Ένωσης, θεσμικού χαρακτήρα εάν για παράδειγμα χρειάζονται νέε αρμοδιότητε, νέα εργαλεία στη διάθεσή του να αποκτήσουν τα εφιστάμενα θεσμικά όργανα, καθώ επίση και τι οικονομικέ και χρηματοπιστωτικέ συνέπειε που θα έχει η όποια απόφαση. Εδώ θα ανέμενε κανείς να επιταχυνθεί η συζήτηση. Από την πλευρά του Συμβουλίου γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τον αντίκτυπο και πιστεύω ότι έχει, θα έχει αξία στη συνάντηση των σχεδόν να συζητήσουμε και εμείς τον αντίκτυπο. Να υπάρξει και στο Κοινοβούλιο λοιπόν συζήτηση για τον αντίκτυπο. Ανάμεσα λοιπόν στα θέματα που είναι τα πιο σημαντικά θα αναφερθώ στις υποπτικές αρχές, το κατά πόσο ο νέο υποπτικός μηχανισμός έχει τα απαιτούμενα εργαλεία στη διάθεσή του, ή θα έπρεπε να έχει περισσότερα. Μετά είναι όλη η συζήτηση για την κεφαλαιακή επάρκεια. Η, η κυρία Μπερές αναφέρθηκε στην ε, ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού την προηγούμενη φορά, ότι θα πρέπει να το ε, εξετάσουμε, παρόλο που δεν είναι, ε, είναι ένα τεχνικό θέμα αλλά ίσως θα έπρεπε επίσης να τεθεί προοδευτικά. όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης και με τη χρηματοδότηση. Μπέιλιν. Με ίδια μέσα δηλαδή. Επίσης το πτωχευτικό δίκαιο και το ερώτημα κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να μας κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση για το πτωχευτικό δίκαιο στο μέλλον. Επίσης η οδηγία που θεσπίζει το πλαίσιο για την ανακάψη και εξηγίαση των πιστοτικών ιδρυμάτων και εδώ έχουμε ερωτηματικά. Και τέλος, ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Μείωση του Ρίσκου αλλά που είναι τα κόκκινα δάνεια. Ένα ζήτημα το οποίο έχει αναδείξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 900 ε, δις. Δεν είναι δυνατό λοιπόν να το αγνοήσουμε. Ένα άλλο θέμα λοιπόν που τίθεται είναι η εφαρμογή των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων θα ήθελαν τα μέλη τη Επιτροπής μας να έχουν περισσότερες πληροφορίες. Πώς λειτουργεί, λειτουργεί στην πράξη. Και τι προβλήματα έχουν παρουσιαστεί, τι δεν λειτουργεί και τι πρέπει να κάνουμε. Επίσης, διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών. Και τέλος το γεγονό ότι την υπέροχη συζήτηση Ορισμένες, κάθε τράπεζα χρησιμοποιεί δικό της σύστημα ε, τήρησης των λογιστικών βιβλίων. Διαφορετικά λογιστικά πρότυπα και ίσως ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα να καταλήξουμε σε διαφορετικές ε, επιλογές όσον αφορά την εξυγένση των στόχος το ε, έκθεσης του, του κειμένου αυτού, του κειμένου εργασίας, είναι να ε, καταλήξουμε σε μια κοινή ε, αξιολόγηση των προγράμματων αυτών, να έχουμε μια κοινή άποψη για το τι ισχύει, ίσως δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Είναι καλύτερα αυτά τα ζητήματα να τα ξεκαθαρίσουμε όταν, τώρα που βρισκόμαστε σε επίπεδο ενός εγγράφου εργασίας, γιατί όταν πλέον φτάσουμε στους νομοθετικούς φακέλους θα υπάρχουν οι συνήθεις διαφωνίες Και το ερώτημα όταν πλέον θα συζητάμε το νομοθετικό φάκελο επίσης θα τίθεται ε, για το πώς ταυτόχρονα θα γίνεται η ε, μείωση του ρίσκου που έχουν αναλάβει οι τράπεζες. Πώς οι δύο αυτές διαδικασίες δηλαδή θα προχωρούν παράλληλα. Αυτό πρέπει να το δούμε πιο μετά. Στο έγγραφο εργασία. Θα ήθελα να ακούσω τις, από τον καθέναν από σας ποιες είναι οι παρατηρήσεις του για το έγγραφο εργασία. Έχω ήδη λάβει σχόλια. Για παράδειγμα από την Ελίζα, ότι και οι τρεις πυλώνες θα πρέπει να είναι ισότιμα, ισότιμοι. Έχω λοιπόν σχόλια τέτοιου τύπου, αλλά αν υπάρχουν και νέα σχόλια για το έγγραφο εργασίας, ευχαρίστως να μου τα εκθέσετε είτε τώρα, είτε γραπτός, ή δυνατόν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην τελική έκδοση του γράφου εργασίας, όπως είχαμε υποσχεθεί, εντός του Μάιου. Ευχαριστώ. Περνάμε στους κοιόδους Η κυρία Φερέρα. πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εστέρ για την παρουσίασή της. Θέλω να επιμείνω σε κάτι που έχω αναφέρει και στο παρελθόν το γεγονός δηλαδή ότι δεν ασχολούμαστε με το περιεχόμενο της νομοθετικής πρότασης που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου πέρυσι, δηλαδή πριν από ένα πεντάμινο. έχουν περάσει ήδη πέντε μήνες και η πρόοδος γίνεται σημειωτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κυρίας Ποια ήταν τα τρία πρωταρχικά σημεία. Θα έλεγα ότι το πρώτο είναι το πιο σημαντικό. Τη θέση των Ευρωπαίων πολιτών και πώς αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τα θεσμικά όργανα. Πώς βλέπουν τα θεσμικά όργανα. έχουμε μια δηλωμένη συμφωνία για τη δημιουργία της ε, Τραπεζικής Ένωσης με τα πρώτα δύο αναγκαστικά βήματα και στο τρίτο έχουμε σταματήσει. Και αρχίζουμε και επεκτηνόμαστε σε, πολύ, άλλα θέματα που είναι με σημαντικά, αλλά ήταν εξίσου σημαντικά και όταν αποφασίσαμε για ένα νέο κανονισμό και για έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, ένα ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης, τότε έπρεπε να μιλήσουμε για τα θέματα, να μιλούσαμε για τα στοιχεία σταθεροποίησης του οικοδομήματος. Τότε έπρεπε από την αρχή να τα συμπεριλάβουμε. Τότε που το κρατικό σύστημα έχασε τον έλεγχο στις τράπεζες. Και είχε συζητηθεί και η νομική βάση στις προηγούμενες φάσεις της συζήτηση. Αναφέρθηκε το άρθρο 114 ως νομική βάση. Τότε το είχαμε λύσει το θέμα και τώρα επανερχόμαστε σε κάτι που είχαμε ήδη ε, διαθετήσει και μάλιστα συνενετικά στο παρελθόν. Το ίδιο ισχύει και για τη διακυβέρνηση. Γιατί το όλο οικοδόμημα ε, φτιάχτηκε για να διαρριχθεί ο δεσμός μεταξύ κράτους και τραπεζών. Και ένα από τα στοιχεία ήταν ε, ένα σταθεροποιητικό στοιχείο στον τραπεζικό τομέα. Και με τη μετάβαση, για τη μετάβαση από ένα εθνικό σύστημα σε μία τραπεζική ένωση στην Ευρωζώνη, η μετάβαση δεν είναι καθόλου εύκολη, είναι πολύ δύσκολη και πριν καν να τεθεί σε ισχύ ε, ο νέος μηχανισμός ε, εξηγή και αρμόδια αρχή, ήδη πυροδοτήθηκε κάποιες ε, έκτακτες δράσεις και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα του Μπέιλιν, γιατί οι χώρες δεν μπόρεσαν να προστατευτούν από το συστημικό αντίκτυπο ενός Μπέιλιν και κυρίως όταν πρόκειται για μικρά ιδρύματα με βάση τα κοινωτικά πρότυπα. Έπρεπε να γίνει με πιο ανοιχτό και ε, τεκμηριωμένο τρόπο, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε, αυξήσουμε την αντίληψη ότι η Τραπεζική Ένωση δημιουργεί ακόμη περισσότερους κινδύνους. Η Έστερ μας παρουσίασε το έγγραφο εργασίας και δεν ξέρω αν ε, θα σχολιάσουμε και την ουσία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά και το περιεχόμενο της πρότασης. Και να διδαχθούμε από τις εθνικές εμπειρίες ό,τι αφορά την προστασία, την εγγύηση των καταθέσεων, να διδαχθούμε από την ε, λειτουργία των IPS, από τη λειτουργία χρόνος, ο χρόνος περνάει. 20 δευτερόλεπτα σου έχουν απομείνει. Α, καλά, τότε τέλος. Όχι, δεν θέλω να σε διακόψω, ολοκλήρωσα. Θα πρέπει να διδαχθούμε από το FTIC, το Μηχανισμό Σταθεροποίησης, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να δούμε τις λεπτομέρειες ε, της πρότασης για το δεσμό των εθνικών συστημάτων εγγύης καταθέσεων, της λειτουργίας, ε, της ταξινόμησης και να διερευνήσουμε τη λειτουργία του άρθρου 11 για να δούμε τις ε, διαφορετικές λειτουργίες των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και τις λειτουργίες, την λειτουργία και την ε, σύνδεση του κοινού μηχανισμού προστασίας για την εγγύηση των καταθέσεων. Πολλές είναι οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίες από την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρότεινα αμέσως μετά την δημόσια κρόαση να επισέλθουμε στο βάθος της ουσίας της πρότασης για να επιταχύνουμε και να διεκπαιρεώσουμε την Τραπεζική Ένωση, τουλάχιστον ως προς τα βασικά της στοιχεία. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχα ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με την προσέγγιση της συγγετρίας και πριν αρχίσουμε να τρώμε θα πρέπει να δούμε ε, το σιτηρέσιο ποιο είναι. Τι προβλέπει το μενού και περιμένω το έγγραφο εργασία με μεγάλη ανυπομονησία. Και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αλλά η πραγματική έναρξη των συζητήσεων θα γίνει όταν λάβουμε το έγγραφο εργασία. Για να δούμε τι εμπίπτει και τι εκπίπτει από το πεδίο εφαρμογή. Τότε μόνο θα ξεκινήσουμε την πραγματική συζήτηση. Το Φεβρουάριο, την τελευταία φορά που μίλησα για το θέμα αυτό, μίλησα ότι είναι κρίμα που δεν έχουμε μελέτη επιπτώσεων και χαίρομαι που το αναφέρει και η συγκεντρία στην εισαγωγή. Γιατί μερικά θέματα έχουν μείνει αναπάντητα ακόμη, δεν έχουν επιληθεί. Επίσης, μείωση του κινδύνου και ρόλος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φυσικά, τα μέτρα μείωση του κινδύνου χρειάζονται, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τέτοια μέτρα μείωση κινδύνου, γιατί ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από τη χρηματοπιστωτική κρίση, τουλάχιστον τελείω. Και πολλές σημαντικές τράπεζε και πολλά κράτη είναι υπερχρεωμένα. Δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε εκτός της συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αγγλική Καταθέσεων. Επίση, να ξαναπώ αυτό που είχα πει και στο παρελθόν. Αν ζητήσουμε από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τράπεζες, ε, τις βόρειες ευρωπαϊκές τράπεζες να σώσουν ε, τους νότιους καταθέτες, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα αυτές, αυτές τις καταθέσεις και να δούμε τι χαρακτηριστικά έχουν. Γιατί όλοι εμείς οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτε μας τους καταθέτες στις χώρες μας θα έχουν την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη κάλυψη και την καλύτερη δυνατή κάλυψη σε περίπτωση που χρεοκοπήσει μια τράπεζα ή μπει σε διαδικασία εξυγίασης. Και θα πρέπει να συμφιλιώσουμε αυτές τις διαφορές μεταξύ των εθνικών τραπεζικών συστημάτων και των διαφορετικών επιπέδων κινδύνων στα συστήματα αυτά. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της δικαιοσύνης που αναφέρατε στην εισαγωγή σας κύριε Και εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ιδέα της δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αγγής Καταθέσεων θα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα δίκαιο. Κάτι που δεν ε, προκύπτει πλήρως ακόμη από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να το δούμε ε, διεξοδικότερα. Και όταν μιλώ για δίκαιο σύστημα εννοώ ότι ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύης καταθέσεων δεν πρέπει να υποβαθμίζει την προστασία που ήδη υπάρχει από τα εθνικά συστήματα εγγύης καταθέσεων. Δεν μπορεί να οδηγήσει ηθικό κίνδυνο, ούτε μπορεί να είναι άδικο στην κατανομή του, των βαρών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και μια τράπεζα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης Καταθέσεων θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια αφετηρία. Θα πρέπει όλα να βρίσκονται στην ίδια αφετηρία και να δούμε και τα, τους του. αν είναι καθαροί όχι. Επίσης, ε, το κόστος ε, παρακαταθήκης legacy cost. Ε, πολλές από τις τράπεζές μας εξακολουθούν να έχουν προβλήματα ε, γιατί φέρουν το κόστος του παρελθόντος της πλάτες τους. Τους έχουν μείνει παρακαταθήκες τέτοιες, τέτοια βάρη, τέτοιες ευθύνες και μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πάντως συμφωνώ ότι θα πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να στρωθούμε στη δουλειά, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα όντως δίκαιο, δίκαιο για όλους τους Ευρωπαίους καταθέτες. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να αναφέρω και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν αρμόδια για, τον, για την συνολική αξιολόγηση του 2014. θα πρέπει να αναλύσουμε αν όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στην ίδια αφετηρία. Θα πρέπει να αποφύγουμε ε, στην ίδια περίπτωση η ECB να είναι και δικαστής και διάδικος. Δεν μπορεί να παίζει κανείς σε δύο ταμπλό ταυτόχρονα. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερος. Όπως είπα, το πραγματικό σημείο φετηρίας θα είναι η υποβολή του γράφου εργασίας. Το περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά το έργο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Εστέρ για την παρουσίαση. Θα σταθώ σε συντομία σε μερικά σημεία. Πιστεύω ότι το θέμα του χρονισμού είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε αρκετό χρόνο για να ξεκινήσουμε τις εργασίες σε αυτό το περίπλοκο ζήτημα, αλλά είναι καιρός να προχωρήσουμε. Επίσης, κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η έκβαση του Βρετανικού Δημοψηφίσματος 23 Ιουνίου και μπορούμε να ξαναμπούμε σε νέα εποχή διαταράξεων και αστάθειας και όταν έχουμε τέτοιο, τέτοια βεβαιότητα μπροστά μας, ε, σίγουρα θα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας. Επίσης, το 2017, σε πολλά κράτη-μέλη και στις κάτω χώρες, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία, στη Γερμανία, επίσης, θα βρεθούμε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε θα έχουμε και το φθινόπωρο το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Πολλές αιστείες ε, έντασης, λοιπόν. Οπότε, αν ε, αφιερώσουμε πολύ χρόνο για την εμβάνθηση, ωραία, δεν έχω αντίρρηση, αλλά γιατί είναι όντω περίπλοκα τα θέματα και χρήζουν εμβάθυνση, αλλά να μην δίνουμε την εντύπωση ότι περιμένουμε για λόγου τακτικής και αφήνουμε το χρόνο να περνά. Επίσης θέλω και την γνώμη της Ευρωπαϊκής, Κεντρική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε τις εθνικές σημαίες, τα εθνικά λάβαρα, γιατί η προστασία των εγγυητών, των καταθετών, συγγνώμη, ε, δεν είναι ανησυχία και προβληματισμός μιας μόνο χώρας. Όλες οι χώρες θέλουν να προστατεύσουν τους καταθέτες τους. Και το να μην έχουμε, να έχουμε σε ορισμένες χώρε πολλά με εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτό θίγει όλου. Ε, δεν θα πρέπει να ε, οχυρωνόμαστε πίσω από εθνικέ θέσεις και συμφέροντα, γιατί η Τραπεζική Ένωση την ζητούσαμε όλοι. Επίσης, το σωρευτικό αποτέλεσμα ε, της ε, ενίσχυσης ε, του Ταμείου Εξυγίασης. Τι θα συμβεί μεταξύ της Τραπεζικής Ένωσης και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όπως επανειλημμένως είπε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρειαζόμαστε ένα σύστημα υγιής καταθέσεων ή ένα backstop, ένα μηχανισμό προστασίας. Γιατί εκεί δεν νομίζω υπάρχει σαφήνεια. Νομίζω πολύ γρήγορα αφήσαμε κατά μέρο το θέμα του μηχανισμού προστασία και του Ταμείου Εξυγίαση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχετικά γρήγορα και με ξυπνάδα για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Και δεν είναι αυτό προϋπόθεση. Πρέπει να γίνονται εκ αυτά τα δύο θέματα. Αν μη τι άλλο για να βρούμε λύση και να συμφωνήσουμε μεταξύ μα. Επίση, να συζητήσουμε και με του επόπτε, τι εποπτικέ αρχέ. Γιατί ένας Ευρωπαίος επόπτης που ε, ελέγχει τις μεγάλες τράπεζες και υπάρχουν και οι ε, εθνικοί επόπτες ε, που είναι αρμόδιοι για τις πιο μικρές τράπεζες. Πώς θα, συνδυάσουμε τους ελέγχους και των δύο φορέων και τι, ποιες είναι οι συνέπειες για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Επίσης, το θέμα της μετάβασης από τη μία στην άλλη φάση. Αν συσσωρεύσουμε πολλά πράγματα, θα τα καταφέρουμε. Αλλά είμαι στη διάθεση της ηγετρίας που φαίνεται ότι επιθυμεί να προχωρήσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ, Σιλβί. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι συμφωνώ απολύτως με την ε, Σιλβί Γκουλάρ ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Η όλη η συζήτηση έχει πάει αρκετά πίσω και έχω αρχίσει πια να αισθάνομαι ότι ορισμένοι επιδιώκουν περαιτέρω καθυστερήσεις και κολυσιέργεια. Και θέλω να πω καθαρά τη γνώμη μου ότι κάθε βήμα αναβολής περαιτέρω μας αφήνει περισσότερο εκτεθειμένους σε συστημικά σοκ. Έχουμε μια πρόταση νομοθετική από τον Νοέμβριο από την Κομισιόν έχουμε ένα σχέδιο τραπεζικής ενοποίησης προσδιορισμένο εδώ και χρόνια με τρεις πυλώνες. Έχουν προχωρήσει οι δύο. Υπάρχει ένας εδώ μέσα σε όποια πολιτική ομάδα και αν ανήκει που να πιστεύει ότι χωρίς τον τρίτο πυλώνα θα έχουμε μια λειτουργική τραπεζική ενοποίηση. Όλα αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν από την εισηγήτρια είναι ερωτήματα που αφορούν μόνο στον τρίτο πυλώνα και όχι στους άλλους δύο. Μήπως παίζουμε εδώ πέρα το παιχνίδι της υποταγής σε ορισμένες εθνικές σκοπιμότητες. Η γνώμη μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η οχύρωση πίσω από εθνικά συμφέροντα και εθνικές σκοπιμότητες αυτή την ώρα είναι καταστροφική για όποιον θέλει να υπηρετήσει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενοποίησης, το οποίο έχει τρεις πυλώνες. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι η τρίτη φορά που συζητάμε και η συγγήτριά μας η κυρία Ντελάνγκη έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά ακόμη εγώ δεν έχω ακούσει τη γνώμη της συγγήτριας. Η πρόταση της Κομισιόν κατά τη γνώμη της κινείται σε θετική κατεύθυνση. Η δική μου γνώμη είναι ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και ότι πρέπει να δούμε, επειδή το θέμα είναι σοβαρό, πώς θα προχωρήσουν παράλληλα και η μείωση του κινδύνου και η αμοιβαιοποίηση του κινδύνου, διότι πρέπει αυτά τα πράγματα να λειτουργήσουν συνδυαστικά. Υπάρχουν ήδη μελέτες, λόμπι που γίνεται από το τραπεζικό σύστημα κρατών μελών, παραδείγματος χάρη της Γερμανίας, κύριε Λούκε, που θέλουν να πούν ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι επικίνδυνη. Πρέπει να την καθυστερήσουμε, πρέπει να μην γίνει ποτέ. Θα το συζητήσουμε αυτό ή θα κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Η πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε, πρέπει να οργανώσουμε μια συζήτηση με την Επιτροπή και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην περιμένουμε να δούμε προς τα που θα φυσήξει ο άνεμος στο Συμβούλιο και να δούμε επιτέλους αυτό το κείμενο εργασίας. Εγώ ακούγοντας την εισηγήτρια να μιλάει τόσο πολύ για το κείμενο εργασίας, κάποια στιγμή παραξενεύτηκα. Λέω, έχει σταλεί κάποιο κείμενο εργασίας το οποίο δεν έχω πάρει. Ας έρθει επιτέλους αυτό το κείμενο εργασίας. Είναι μήνες που η εισηγήτρια έχει αναλάβει την ε, εντολή. Έχουμε κάνει και συνάντηση σκιωδών εισηγητών. Της δώσαμε και την άνεση να παρουσιάσει την πρότασή της μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, όταν θα μπορούσε να έρθει και νωρίτερα, αλλά για να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και όχι για να ροκανίζουμε το χρόνο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ενοποίηση θα πετύχει αλλά με μόνο δύο πυλώνες. Δεν γίνεται. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες αυτή την ώρα. Ζητώ απλώς να επιταχύνουμε, η εισηγήτρια να φέρει κείμενο εργασίας και να ορίσουμε συνεδριάσεις για να συζητήσουμε με την, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της επιτέλους και όχι μόνο τα γύρω-γύρω και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που και αυτή ασφαλώς έχει μια, έναν βαρύνοντα λόγο ε, στην εξέλιξη του θέματος. Ευχαριστώ. Thank you. Now for the Ευχαριστώ. Φίλιπ Λάμπας για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Έστερ συνάδελφοι. Συμφωνώ με, ό, όλους που είπαν ότι πρέπει να, κάτι να κάνουμε, κάτι να καταφέρουμε. Το εγχείρημα δεν είναι να ε, δουλέψουμε προσχηματικά, Πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Ο Δημήτρης είπε ότι η πρόταση της Κομισιόν πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί. Όχι, ε, δεν είναι επειδή δεν υπάρχει ε, εκτίμηση επιπτώσεων που θα την πρέπει να την απορρίψουμε. Υπάρχουν δύο θέματα που μπαίνουν και ξαναμπαίνουν και που κρύβουν την πολιτική βούληση να μην βρούμε αποτέλεσμα. Συχνά ακούω για τους ηθικούς κινδύνους, με την έννοια ότι ναι, αλλά γιατί οι Γερμανοί φορολογούμενοι να ε, πληρώσουν για κακοδιαχειριζόμενες Ιταλικές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ό,τι και να πει κανείς, ε, δεν έχουμε λύσει το θέμα του too big to fail. Είναι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν. Η Deutsche Bank, ε, δηλαδή είναι γερμανική ε, τράπεζα επειδή λέγεται Deutsch, είναι ένα ε, παγκόσμιο hedge fund. Και αν υπάρχουν ε, κίνδυνοι εκεί, βεβαίως θα υπάρχουν και διάφοροι, διάφοροι που θα χάσουν, που δεν είναι μόνο Γερμανοί, επενδύουν σε μια τράπεζα γκανιστερική, αν αποτύχει τότε φέρουν τους κινδύνους. Λογικό είναι. Ε, μην μιλάμε όμως για Γερμανούς φορολογουμένους. Μην λέμε ότι αν η τράπεζα έχει τα κεντρικά της σε μία χώρα, είναι γερμανική ή, ή γερμανοϊταλική ή οτιδήποτε. Αν το πιστεύετε αυτό, να είστε ε, έντιμοι και να μας βοηθήσετε να βάλουμε τέλος στο σύνδρομο του big to fail. Δεύτερον, λέμε ας πούμε ότι έχουμε υπερβολική έκθεση στο δημόσιο χρέος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, όντως. Νομίζω όμως ότι όποιοι μελετήσουν το θέμα προσεκτικά θα δουν ότι το θέμα αφορά τη συγκέντρωση, τη συγκέντρωση οποιοδήποτε κινδύνου αλλά και συγκεκριμένου κρατικού κινδύνου. Μια τράπεζα δηλαδή μπορεί να έχει εκτεθειμένο μεγάλο κεφάλαιό της σε δημόσιο χρέος, αν όμως είναι από πολλές χώρες, ας πούμε ένα καλάθι χωρών της Ευρωζώνης που σταθμίζεται ε, σύμφωνα με το βάρος της κάθε χώρας και φανταστείτε η ελληνική συνιστός αυτού του χρέους θα θεωρείται πιο επικίνδυνη, αλλά αυτή θα αντισταθμιζόταν από λιγότερη, ε, λιγότερο επικίνδυνη ε, ε, αξιολόγηση του γερμανικού ιταλικού κινδύνου. Στο βαθμό που διαφοροποιείς το καλάθι και λες ότι οι ιταλικές τράπεζες δεν είναι πολύ εκτεθειμένες στο ιταλικό χρέος ή οι βελγικές στο βελγικό χρέος κλπ. Στο βαθμό που υπάρχει διαφοροποίηση είμαστε ασφαλείς. Και αυτό με ε, φέρνει στο εξής. Ορισμένοι θεωρούν το επιχείρημα μείωση του χρέους ως πρόσχημα για να μην γίνει δουλειά. Δεν λέω ότι αυτό είναι ε, η πρόθεσή τους, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί εδώ. Και εκεί μπορεί να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με τη Σιλβή, θα το δούμε αυτό. Εδώ έχουμε δύο παράλληλες οδούς που για μένα όμως συνδέονται. Πρέπει ή μάλλον αντί να πούμε δεν θα κάνουμε τίποτα, συνεχίζουμε, προχωρούμε παράλληλα και στα δύο. Άρα συμφωνούμε να βεβαιωθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, γιατί ε, επειδή από τότε που κάναμε BRD ε, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα υπάρχουν κενά στο δίχτυ μας. Αν μπορούμε το εγχείρημα αυτό να το ε, αξιοποιήσουμε για να κλείσουμε κάποια κενά, ας το κάνουμε και εκείνοι που θέλουν να ε, καθυστερήσουν την υπόθεση του ΕΣΑΚ ε, θα βρεθούν σε ε, μειονεκτική θέση γιατί εμείς θα δώσουμε συνολική λύση. Βεβαίως και εγώ περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω το έγγραφο εργασίας για να αρχίσουμε την αντιπαράθεσή μας και να καταλήξουμε πιστεύω σε μια καλή συμβιβαστική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρκο Ευχαριστώ. Εν συντομία θα επαναλάβω κάποια σημεία που ήδη ανέφερα και στις προηγούμενες συζητήσεις. Και εγώ περιμένω με ανυπομονησία το έγγραφο εργασίας για να έχουμε πιο σαφείς βάσεις για τη συζήτηση για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε κάτι έχοντας ως βάση κάποια έγγραφα εργασίας. Αυτό περιμένουμε. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Το, τραπεζικό, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα υποφέρει το σύνολο του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος υποφέρει και ταλανίζεται και από εσωτερικά προβλήματα και από δυνητικούς εξωτερικούς κινδύνους. Και αρκετές, αρκετές οφερές ήταν και οι προβλέψεις ε, του Αμερικανικού FDIC, του Federal Reserve και το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για τις πιο σημαντικές και μεγάλες ε, αμερικανικές τράπεζες. Ακόμη και μεγαλύτερη, για παράδειγμα, τράπεζα δεν θα μπορούσε να αντέξει σε πολύ μεγάλο στρες. Οπότε, αν μια τέτοια τράπεζα χτυπηθεί από κρίση, ποια θα ήταν η συνέπεια στο ευρωπαϊκό ε, τραπεζικό σύστημα που ήδη υφίσταται μεγάλες πιέσεις. Είναι λοιπόν ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που όχι μόνο θα δίνει κάποια εχέγγυα ασφάλειας στους καταθέτες, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει μια χρηματοοικονομική σταθερότητα σε ολόκληρο το σύστημα. Και μια και αυτός είναι ο στόχος μας, που είναι και πολύ ευρύς, ε, είναι σημαντικός και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να λειτουργήσει τελικά ο μηχανισμός αυτός. Γιατί αν περιοριστούμε σε ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων, που θα στηρίζεται στις αρχικές προτάσεις που λάβαμε, ένα τέτοιο σύστημα θα είναι ανεπαρκές και δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαραίτητη σταθερότητα. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επεκτείνουμε το έργο μας ώστε να διορθώσουμε κάποιες στρεβλώσεις που δημιούργησαν οι προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις και που βασανίζουν την αγορά. Το bail-in, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για παράδειγμα ε, και το BRRD, το σύστημα εξηγής ανάκαψης τραπεζών. Ακόμη δεν έχουμε διαμορφώσει άποψη. Φαίνεται ότι οι τρέχοντες οργανισμοί που θα υπερβαίνουν ένα ποσό θα εντάσσονται στον υπολογισμό των επενδύσεων. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και ε, στους λογαριασμούς ε, τρεχουσών πληρωμών. ώστε να μένουν χρήματα και εκεί. Αλλά δεν μπορεί να θεωρείται ένας ε, λογαριασμός τρεχουσών πληρωμών επένδυση. Αν έχουμε ένα backstop, ένα μηχανισμό προστασίας και μια εγγύηση στην οποία θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό θα είναι καλό και απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον Φίλιπ Λάμπερτς και ως Ιταλός φορολογούμενος θα ανησυχούσα πολύ αν έπρεπε να σώσω με τα δικά μου χρήματα μια μεγάλη τράπεζα, την Deutsche Bank για παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι το ποστο έκθεσης σε παράγωγα είναι πολύ μεγαλύτερο. Κάτι που ίσως θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα. Και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός ε, θα πρέπει να βαθύνει περισσότερο στα περιουσιακά στοιχεία του επίπεδου 3 και στα παράγωγα, στα οποία είναι εκτεθειμένα κυρίως οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και που δεν εμπίπτουν στο σύστημα clearing. Αυτό είναι επικίνδυνο όμως και ο κίνδυνος ε, που απορρέει τεράστιος. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο στη συζήτηση αυτή είναι το εξής. Με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εγγύης καταθέσεων, για να θωρακίσουμε τις καταθέσεις, δεν θα πρέπει να δεχτούμε ως αντάλλαγμα, ως αντιστάθμισμα, κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του συστήματος αν συμφωνήσουμε σε ένα μηχανισμό για να βελτιώσουμε τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, δεν μπορούμε να δίνουμε ανταλλάγματα που θα την υπονομεύουν. Βέβαια, κάποια κρατικά ομόλογα σίγουρα θα περιέχουν κινδύνους, αλλά δεν θα, θα πρέπει να αποφύγουμε επιζήμια αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Και εγώ περιμένω το έγγραφο εργασίας. Αλλά ως πότε θα περιμένουμε. Ολόκληρες εβδομάδες έχουν περάσει. Ήρθε η ώρα επιτέλους να στρωθούμε στη δουλειά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα έγγραφο εργασίας. Δεν έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις από την τελευταία φορά που το συζητήσαμε. Και τις τελευταίες εβδομάδες διαβάζουμε στις οικονομικές εφημερίδες, για παράδειγμα στην Αυστρία είχαμε τέτοιες ειδήσει ότι ε, έχουν μια τεράστια τρύπα από ό,τι φαίνεται από τους πρώτους υπολογισμούς. 54%. Επίσης, ε, το σύστημα εγγύης καταθέσεων μερικές φορές ε, χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Παρουσιάζεται ως μια τραπεζική ένωση που λέει ότι οι μεγάλες τράπεζες ε, θα πληρώνουν για αυτούς για τις κακές τράπεζες και ακόμη και οι μικροί καταθέτες θα πρέπει να συμμετέχουν στη διάσωση, παρόλο που δεν είναι τα μεγάλα κεφάλαια. Και επίση έχουμε το όριο των καταθέσεων στα 100.000 ή ε, το μύθο ότι ε, θα υπάρξει εγγύηση καταθέσεων και θα αγγίξουμε τους ε, λογαριασμούς ταμιευτήριων, αποταμιεύσεις. Επίσης υπάρχει διαφορά μεταξύ βορρά και νότου. Υπάρχει ένα χάσμα που αυξάνεται όλο και περισσότερο. Ο κύριος Παπαδημούλης θέλει ε, να τα επιταχύνουμε όλα, να καταλήξουμε σωστές αποφάσεις ε, το συντομότερο δυνατό, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη ε, επικρίνουμε εκείνους που συστηματικά πατάν φρένο και επιβραδύνουν τη διαδικασία και Ε, το σχόλιο ότι για να μειώσουμε τον κίνδυνο θα πρέπει να τον αμοιβαιοποιήσουμε. Ένα σταθές όμως ε, ε τραπεζικό σύστημα δεν θα είναι μόνο πρόβλημα των χωρών του Νότου. Ο κίνδυνος αυτός θα επηρεάσει και τις χώρες του Βορρά. Ιδιαίτερα αν το σύστημα καταρρεύσει. Βέβαια δεν μπορούμε να βιάσουμε τα πράγματα και να λάβουμε υπόψη και τις ανησυχίες των χωρών του Βορρά. Και χώρες που έχουν ήδη συστήματα καταθέσεων να μην βρεθούν σε δυσμενή θέση από ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Θα πρέπει να έχουμε ένα δίκαιο σύστημα για το σύνολο της Ευρώπης. Δίκαιο και ισορροπημένο. Παρόλο που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τους κινδύνους. Πιστεύω ότι ακόμη και αν μπορούσαμε να τους υπολογίσουμε, θα καταλαβαίνουμε πολύ σύντομα ότι είναι μεγάλο το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου που περνάει από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Ευχαριστώ. Ε, είχε βγει ένα φυλάδιο από την ΕΚΤ πολύ ενδιαφέρον πριν από λίγο καιρό και αφορούσε τις κρατικές ενισχύσεις και την ποσότητά τους τα τελευταία χρόνια. Και δεν, έβγαινε από εκεί ότι το πρόβλημα δεν επικεντρωνόταν στο Νότο, αλλά αφορούσε περισσότερο το Βορρά. Γιατί υπάρχει η αντίθετη εντύπωση ότι οι νότιες χώρες χρειάζονται πολλές ε, επιδοτήσεις με βάση ε, ιστορικά δεδομένα που όμως αλλάζουν. Πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye, πρώτος ομιλητής. Ο κ. Ζάλμπα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ Εστέρ για την τεράστια προσπάθεια που κάνεις και το δύσκολο έργο σου. Μερικά σύντομα σχόλια. Όλοι συμφωνούμε ότι μια τραπεζική ένωση θα πρέπει να παρτίζεται από τρεις πυλώνες. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο μόνο. Είναι λογικό λοιπόν να συνεχίσουμε τις εργασίες ώστε να συμπεριλάβουμε και τον τρίτο πυλώνα, να τον κάνουμε πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό. Και αν προσθέσουμε σε αυτό και το πολιτικό πλαίσιο που μας εξήγησε η Σιλβή, που δεν είναι το πιο γαλήνιο δυνατό, έχουμε έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουμε τις νομοθετικές εργασίες ως προς την έκθεση Ντελάγκε. Φυσικά συμφωνώ με την εισηγήτρια να αποφύγουμε τους ηθικούς κινδύνους, και αφήνοντας κατά μέρους ε, όλα τα συναισθήματα, τα έντονα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η έκθεση, θα πρέπει να συνδυάσουμε το θέμα των κινδύνων με τα απαραίτητα μέτρα μείωσης ε, ώστε να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, που είναι ο κοινό μας στόχος. Αναφέρθηκε ο δεσμός που υπάρχει στην έκθεση αυτή με άλλες εκθέσεις που επίσης εκπονούμε στην Επιτροπή μας. Όλα είναι αλληλένδετα και αν αυτοί οι δεσμοί ε, χρησιμοποιηθούν για να επιταχυνθούν οι εργασίες και σε άλλες εκθέσεις που εκ παραλλήλου καταρτίζουμε, Πολύ ωραία. Είναι ευπρόσδεκτο και θεάρεστο. Τώρα όμω, αν αυτοί οι δεσμοί, αυτές, αυτοί οι σχετισμοί χρησιμοποιηθούν ω πρόσχημα για να επιβραδύνουμε τι εργασίε, ε, δεν συμφωνώ. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτέ οι σχέσει μεταξύ των διαφόρων εκθέσεων για να εχμαλωτήσουμε αυτή την έκθεση και να την κρατήσουμε όμοιρο της εξέλιξης άλλων εκθέσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να επιταχύνουμε τις εργασίες. Ευχαριστώ ο Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε μία από τις σημαντικότερες συζητήσεις της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας. Και λέω της παρούσας γιατί φαίνεται ότι υπάρχει και μία διάθεση για να μην επιταχύνουμε τη συζήτηση και να μην διεκπαιρώσουμε γρήγορα τι εργασίε. Μπορούμε να συζητούμε αν αρκεί ή όχι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύηση Καταθέσεων για να συμπληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και το, για το αν χρειάζονται συμπληρωματικά μέτρα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει σαφής πλειοψηφία υπέρ της άποψη ότι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύηση Καταθέσεων εκ των όνων ουκάνευ προπόθεση, απαραίτητη προπόθεση και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να το συζητήσουμε το συντομότερο δυνατό. Αυτή τη στιγμή ακούμε πολλά για το πιθανό ηθικό κίνδυνο του νέου ευρωπαϊκού συστήματος. Το θέμα του ηθικού κινδύνου θα το βρούμε μπροστά μας και στο μέλλον. Με, τον επιμερισμό των ευθυνών και τα, τα κίνητρα που θα δοθούν και στον εποπτικό μηχανισμό. Και από τη στιγμή που θα περικοδοτήσουμε πλήρως το Ταμείο Εξηγήσει, θα έχουμε έναν ενίο εποπτικό μηχανισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το θέμα όμως ε, ε της εγγύησης των καταθέσεων ε, θα εποπτεύεται σε εθνικό επίπεδο. Οπότε ο επόπτης δεν θα διαχειρίζεται τις εγγύησεις καταθέσεων και αυτός που θα διαχειρίζεται τις εγγύησεις καταθέσεων εθνικά, ποιος θα τους ε, εποπτεύει. Υπάρχει μια ισορροπία λοιπόν μεταξύ του ηθήνοντος που λαμβάνει τις αποφάσεις και του επόπτη και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί με το σύστημα αυτό. Τώρα, αναφέρθηκαν διάφορα συμπληρωματικά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. Αναφέρθηκε η συζήτηση για το δημόσιο χρέος. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και μία, δεν ξέρω αν πρέπει να σκεφτούμε μία αποκλειστική ρυθμίση για τα κράτη-μέλη της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Κάτι τέτοιο όμως θα δημιουργούσε μεγάλες ε, διακρίσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και της Τραπεζικής Ένωσης και των υπολείπων. Και από τη στιγμή που θέλουμε και χρειαζόμαστε ενιαία χρηματοοικονομική αγορά και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τις προτάσεις για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, θα ήταν ε, επιζήμιο να έχουμε διαφορές μεταξύ χωρών εντός και εκτός της Τραπεζικής Ένωσης. Επίσης, πού οφείλεται το δημόσιο χρέο και η κρίση του δημόσιου χρέου ποια είναι τα αιτιά του. Γιατί μας έπεσε στο κεφάλι να ανακατεύεται και δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να ε, περιορίσουμε την έκθεση των τραπεζών στο δημόσιο χρέος. Νομίζω ότι με εξαίρεση την Ελλάδα η κρίση του δημόσιου χρέους οφείλεται στην έλλειψη της Τραπεζικής Ένωσης. Γιατί όταν μπήκαμε στην κρίση δεν είχαμε Τραπεζική Ένωση. Αν είχαμε τραπεζική, επειδή δεν είχαμε Τραπεζική Ένωση, τα, τα κράτη με το προπολογισμό του προσπάθησαν να σώσουν, να αντιμετωπίσουν την κρίση των τραπεζών και αυτό δημιούργησε δημόσιο χρέο. Οπότε δεν θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τέτοιε κρίσει δημόσιου χρέου με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε τώρα. Αν είχαμε τραπεζική ένωση θα είχαμε πολύ λιγότερη κρίση δημόσιου χρέου. Επίση θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση ε, με το legacy debt, αυτή το, το βάρος του παρελθόντος, τα χρέη του παρελθόντος, ώστε το νέο σύστημα να μην καταρρεύσει εξαιτία του βάρους του παρελθόντος. Και επίσης να έχουμε και περιοσιακά στοιχεία απαλλαγμένα από κίνδυνο. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν θα πρέπει να εξεταστούν. Ευχαριστώ. Η Ντανίτα Χίμπνερ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω κι εγώ δύο λόγια για αυτό που η Έστερ το είπε η πλευρά των καταθετών. Συμφωνώ μαζί της, δεν ξέρουμε πολλά σχετικά με το πώς δημιουργούν τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Ξέρουμε όμως ότι χρειάζεται εναρμόνιση πριν θεσπιστεί το ΕΣΑΚ και θα πρέπει να συμφωνήσουν, να αποφασίσουν οι εμπλεκόμενοι αν η εναρμόνιση θα γίνει πριν αρχίσουμε να συνενώνουμε τους σπόρους ή αν θα γίνει παράλληλα. Επίσης πιστεύω ότι η εναρμόνιση αυτή θα είναι μια πρόκληση όταν πρόκειται για τις εθνικές επιλογές, διακριτικές ευχέρειες, ιδιαίτερα όταν σκεφτόμαστε το επίπεδο το κάλυψης, τη διάρκεια της κάλυψης και την επιλεξιμότητα των εγγυήσεων ε, γενικότερα. Υπάρχει και μια αναντιστοιχία μεταξύ του ΕΣΑΚ και των εθνικών συστημάτων όταν πρόκειται για το επίπεδο στόχο της ε, κάλυψης. Επίσης ένα μεγάλο θέμα σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια είναι τα εναλλακτικά μέτρα. Πάλι υπάρχουν χώρες που ε, προχωρούν τον κανονισμό προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα, ε, στο ΕΣΑΚ δεν, δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα. Μια ερώτηση προς την Κομισιόν Νομικής Φύσεως. Το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει άμεση ε, μεταφορά ε, συνεισφορών από τα εθνικά ταμεία στα ε, συστήματα εγγύησης θα χρειαστεί, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται διακυβερνητική ε, συμφωνία για τη μεταφορά των κονδυλίων και επίσης τις πιστώσεις ε, πληρωμών που δεν αναφέρονται στην πρόταση για το ΕΣΑΚ ενώ έχουν γίνει δεκτές ως συνεισφορές στα ΣΕΚ και στα, εθνικά δηλαδή συστήματα εγγύησης. Ποιο είναι το σκεπτικό της παράβλεψης αυτής και ποια θα ήταν τα υπέρ και τα κατά ενδεχομένως ε, στο να μπορεί να προβλέπετε κάτι τέτοιο και στα πλαίσια του ΕΣΑΚ. Ευχαριστώ. Κώστας Μαυρίδης. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζω με ένα βασικό ερώτημα. Γιατί χρειάστηκε η Τραπεζική Ένωση και θα δώσω μια απάντηση που θα βρει νομίζω σύμφωνους όλους. Ότι αυτή ήταν η αντίδρασή μας, η ευρωπαϊκή απόκριση στην χρηματοπιστωτική κρίση με στόχο να ξεχωρίσουμε τις τράπεζες από τον κρατικό τομέα, το δημόσιο. Νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν ο πρώτος στόχος. Και Έτσι, εργαζόμενοι με ε, συνέπεια, καταλήξαμε στην ε, αρχιτεκτονική της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Βέβαια, πολλές φορές, ως επιτοπλίστων, η ηθική και η πολιτική δεν πάνε μαζί. Οπότε, ξαναρωτώ, πώς ξέρουμε από την αρχή ότι πώς το ξέραμε από την αρχή ότι ο τρίτος πυλώνας ή ότι οποιοδήποτε πυλώνας δεν θα αφορμοζόταν. Αν ισχύει αυτό, τότε οι άλλοι δύο πυλώνες δεν θα ήταν οι ίδιοι. Σήμερα το πρωί παρακολούθησα τη γερμανική συζήτηση για την εγγύηση των καταθέσεων και δεν εκπλήσωμε ότι κάποια επιχειρήματα μεταφέρθηκαν σε αυτή τη συζήτηση 100% τα ίδια. Εντάξει, κατανοητό μεν, αλλά πιστεύω ότι όταν κάναμε τη συζήτηση αυτή πριν από λίγους μήνες, κάποια, ε, ετέθησαν κάποια θέματα τεχνικής φύσεως. Τώρα έγιναν 5-6. Από δύο μήνες, σε δύο μήνες χρόνο θα γίνουν 10 ή 20. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι θέλουμε την Τραπεζική Ένωση... Ε, στο πνεύμα στο οποίο είχαμε συγκλίνει από την αρχή ή δεν τη θέλουμε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με δύο ακόμα σύντομα σχόλια. Ο ηθικός κίνδυνος. Εγώ ήμουν στο δημόσιο πολλά χρόνια. Α, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες ήμουν πολλά χρόνια. Αν θέλει κάποιος εγγύηση καταθέσεων με μηδενικό ηθικό κίνδυνο, εγώ μπορώ να σας πω ε, ότι ε, ως ε, ότι ε, αυτός που το λέει αυτό δεν θέλει εγγύηση καταθέσεων. Δεύτερον, τώρα που μιλάμε, ε, σίγουρα γίνονται διακρίσεις κατά, ε, μεταξύ των και κατά των καταθετών ακόμα και εκείνοι από εμάς που ανησυχούμε και θέλουμε να έχουμε ίσους όρους του παιχνιδιού μεταξύ ιδιωτικών εταιριών και ιδιωτικών τραπεζών και εκεί δεν είναι ίσοι οι όροι του παιχνιδιού. Ξέρουμε ότι οι τράπεζες ε, υποφέρουν ε, στα πλαίσια τα τωρινά. Ευχαριστώ, Μίχαλ Σόγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην υπάρξει διχασμός μεταξύ της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω σαφή διχασμό όπως ισχυρίζονται κάποιοι μεταξύ Βορρά και Νότου. Είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη εικόνα και πρέπει να τη δούμε με πιο διαφοροποιημένο τρόπο. Στις ευρωπαϊκές συνθήκες έχουμε τις αρχές της ε, αναλογικότητας και της επικουρικότητας και ένα μεγάλο ερώτημα από τη δική μου την πλευρά είναι το εξής. Ήδη έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα εγγύησης των αποταμιεύσεων του κόσμου, αλλά δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε γιατί πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η υλοποίηση. Επειδή κάποια κράτη-μέλη δεν θέλουν να εφαρμόσουν το ισχύον σύστημα ή επειδή δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Αν απαντηθεί, ίσως δεν υπάρχει ε, όφελος από, τον από το ΕΣΑΚ δεν θα δώσει κάτι παραπάνω. Το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το ανταγωνιστικό πλαίσιο. Εγώ σοκαρίστηκα όταν διάβασα πρόσφατα σε γερμανική εφημερίδα ότι οι μεγάλες ιδιωτικές ε, τράπεζες στη Γερμανία, η Commerzbank και η Deutsche Bank δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν πλέον ε, ε, ε, ε, και δεν θέλουν δηλαδή να είναι αλληλέγγυες με τις ε, μικρές τράπεζες. Υπάρχει ένα όριο πάνω από 100.000 για την εγγύηση. Οπότε η εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης των 100.000 ήδη αλλάζει πλέον το ανταγωνιστικό πλαίσιο στις μερικές αγορές. αν το σύστημα το προτείνουμε, όπως το λέει η Κομισιόν, αλλάζει για κάποιες τράπεζες το ανταγωνιστικό πλαίσιο. Και είχαμε πρόσφατα και μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο Γκέτε της Φραγκφούρτης που λένε ότι υπάρχουν πλέον επιστημονικά πορίσματα που δείχνουν ότι το ρυθμιστικό μας πλαίσιο κάνει διακρίσεις σε βάρος των μικρών και μεσαίων τραπεζών. Άρα πρέπει να γίνει εκτίμηση επιπτώσεων όλων αυτών, γιατί δεν είναι δυνατόν το ρυθμιστικό πλαίσιο να ε, δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των μικρομεσαίων τραπεζών, όπου και να βρίσκονται. Δεν ε, έχει σημασία η χώρα. Πρέπει όμως ε, να είναι ίση η ανταγωνιστική όρη του παιχνιδιού. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, ο κύριος Λούκε. Πολλοί ομιλητές είπαν ότι, συμφωνούν, ε, ε, συμφωνούμε όλοι ότι, ε, σχετικά με τον τρίτο πυλώνα. Εγώ δεν τον θέλω τον τρίτο πυλώνα των τραπεζών, άρα δεν συμφωνούμε όλοι και κατάλαβα ότι και ο κύριος Τόιρε ε, δεν έχει πιστεί για την αναγκαιότητα του τρίτου πυλώνα τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν εδώ υπέρ του ΕΣΑΚ δεν είναι καθόλου πιστικά, κάθε άλλο. Ο, κύριος, ο Κώστας Μαυρίδης είπε ότι το αρχικό ε, κίνητρο ήταν ε, το, τον κίνδυνο του κρατικού χρέους ε, να το διαχωρίσουμε από το κίνδυνο του χρηματοοικονομικού τομέα. Ε, ο Φίλιπ Λάμπερτς το ανέφερε αυτό όμως και είπε ότι καμία τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να διατηρεί μόνο κρατικά ομόλογα της δικής χώρας. Μπορεί να πιεστεί ρυθμιστικά, αλλά δεν, δεν, δεν είναι υποχρεωμένη καταρχήν. Ε, μπορεί να γίνει διαφοροποίηση του κινδύνου με ανάλογο χαρτοφυλάκιο ε, και λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμιση των χωρών σε σχέση με τον κίνδυνο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτό να είναι επαρκής αιτιολόγηση του τρίτου πυλώνα. Μετά, προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε το θέμα του ηθικού ε, κινδύνου. Και αυτό είναι λάθος, γιατί αυτό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα του ΕΣΑΚ και του τρίτου πυλώνα, ότι έχουν ε, δημιουργηθεί πολλά ε, κίνητρα στα πλαίσια του μικρού κινδύνου. Στα πλαίσια της ευρωκρίσης το 2010 πολλοί ισχυρίστηκαν, δεν συμφωνώ απόλυτα αλλά αναφέρομαι σε αυτούς, ε, σε είναι γνωστή, πολλοί είπαν ότι η υπερχρέωση στις ε, νότιες χώρες του ευρώ ε, δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων διότι είχε υπάρξει έμεσα πρόβλεψη του bailout, δηλαδή έπαιξε ρόλο ο ηθικός κίνδυνος εδώ. Και βέβαια θα επαναληφθεί αυτό εάν δεχτούμε τον τρίτο πυλώνα στην Τραπεζική Ένωση, γιατί ε, στην οικονομική πολιτική λαμβάνει την υπόψη η κερδοφορία των εταιριών ε, και αυτό επηρεάζει βέβαια και την κερδοφορία των τραπεζών. Ε, οι κυβερνήσεις θα έμπαιναν λοιπόν στον πειρασμό να αναλάβουν υψηλούς κινδύνους αν θεωρούσαν ότι διασφαλίζονται με την συνένωση του κινδύνου. Ε, νομίζω λοιπόν ότι το σωστό, η σωστή απάντηση είναι ότι στο βαθμό που ε, τα, τα, τα κράτη-μέλη έχουν την οικονομική την οικονομική τους ε, πολιτικής θα πρέπει να έχουν και τα ΣΕΚ τους ε, και περιτεύει η θέσπιση ενός ΣΑΚ γι' αυτό το λόγο. Ευχαριστώ. Και τώρα η συγγήτρια. Σα ευχαριστώ. Πράγματι, ακούγοντα και τους τελευταίους δύο ομιλητέ έχουμε το σύνολο των απόψεων που έχουν ακούσει για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων και για αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά, όπως είπε και η κυρία Φερνάντε. Ε, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο, με το οποίο συμφωνούμε περισσότεροι, ίσως όχι ο κύριο Λούκε, όχι κάποιοι άλλοι, είναι να δούμε ποιε είναι οι συνθήκε υπό τι οποίε ο Έντι στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλεια Καταθέσεων, θα μπορούσε να επιτύχει. Και τότε θα πρέπει να το υλοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε ε, χωρίς συζήτηση ναι γιατί το υποσχεθήκαμε ή όχι γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είχα προτείνει στους συναδέλφους να έχουμε ένα κείμενο εργασίας το οποίο θα ε, καταγράφει επακριβώς ποιες θα είναι οι συνθήκες, οι ε, προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σωστά ο έντις. Και χαίρομαι λοιπόν για την ε, παρέμβαση σε σχέση με το δημόσιο ρίσκο το, η στάθμιση του ρίσκου θα πρέπει να γίνεται διαφορετικά ανάλογα με την προέλευση του χρέους, για παράδειγμα. Τέτοιες προτάσεις με βοηθούν να αντιμετωπίσω τα ζητήματα. Δεν με βοηθεί μια προσέγγιση που λέει θα ήθελα να το είχα χτες, ότι θα έπρεπε να βιαστούμε. Ούτε επίσης με βοηθάει ένα, μια ξεκαθαρή ε, άρνηση το ίδιο επίση δεν με βοηθάει να υποστηρίζουμε ότι μπορούμε να εξαναγκάσουμε τους Γερμανούς. Τι να κάνουμε. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια πρόταση την οποία να μπορούν να την υποστηρίξουν οι περισσότεροι. Και για να συμβεί αυτό πιστεύω ότι ε, η πρόταση πρέπει να έχει τις σωστές προϋποθέσεις και αυτές που ανέφερε ο κ. Στόιρερ και άλλοι. Γιατί χρειάζεται υποστήριξη των κρατών μελών. έχουμε ήδη δεχτεί ότι δεν υπάρχουν καταθέτες ή πιστωτές πολλών ταχυτήτων. Επομένως, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα θέσει τα κράτη-μέλη, ορισμένα από τα κράτη-μέλη, σε μια κατάσταση δυσχερέστερη από την οποία ξεκίνησαν, από την οποία βρίσκονται τώρα. Το ερώτημα λοιπόν που έθεσε και ο κ. Στοέρε είναι το ε, εξή. Εάν κάποιος έχει βάλει τα χρήματά του σε μια τράπεζα η οποία δεν έχει διασυνοριακέ συναλλαγέ. Έχει μικρό ποσοστό διαχείριση συνοριακών συναλλαγών. Και το έκανε αυτό επί τη βάση τη πίστη. Αυτέ ε, είναι σε μια διαφορετική κατηγορία. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα αναλογικότητα. Το θέλει, θέτει ο κύριο Τόιρερ και το θέτουν και άλλοι. Ε, παρόλο που ίσω κάποιοι συνάδελφοι να το θεωρούν ε, αστείο, είναι ουσιαστικό γιατί ορισμένοι από αυτού του καταθέτε το γεγονό ότι έχουν ε, μία ε, προστασία των 100.000 ευρώ μπορεί να τους το εξασφαλίσει και η πρώτη φάση του έντις. Δεν λέω ότι εγώ την προτιμώ αυτήν την κατάσταση, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Επίσης, το ζήτημα που έθιξε η κυρία Φερνάντες. Ποια είναι η σχέση των μεγάλων συστημικών τραπεζών με τον, τις πολυάριθμες μικρότερες τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν τέτοιου τύπου έκθεση. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει στις μεγάλες τράπεζες, στους μεγάλους παίκτες. Και κατά τα άλλα θεωρούν ότι η εποπτεία σε εθνικό επίπεδο των μικρότερων τραπεζών μπορούμε να ε, ε, ε, θεωρήσουμε απριόριο ότι λειτουργεί. Άλλο ένα ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε. Υπάρχουν και άλλα πολλά, κύριε Πρόεδρε. Και Χαίρομαι που ορισμένοι από τους συναδέλφους απάντησαν στις ερωτήσεις που είχαν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις μας. Δηλαδή, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να αναλάβουμε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πώς πρέπει να δομήσουμε τελικά το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Προς την κυρία Φερέιρα. Μάλιστα. Εάν θέλετε να δείτε στα γρήγορα αυτό το έγγραφο εργασία, γιατί θεωρώ ότι και εσεί όπω και άλλοι συναδελφοί είστε από αυτού που το θέλουν να το δουν στα γρήγορα. Δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρέπει το, το, το, έγγραφο εργασία πρέπει να καταγράφει τι ορθέ προποθέσει. Εν πάση περιπτώσει. Εάν αυτό πιστεύετε, εγώ θα κάνω απλώ παραπομπέ στην πρόταση τη ΕΔΙΣ, στην πρόταση τη Κομισιόν, συγγνώμη για τον ΕΔΙΣ, και ε, στην εφιστάμενη νομοθεσία. Αλλά και τότε πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συζητήσω τη συνεργασία σα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι απλώ κάποιο να μου ζητάει να παρουσιάσω το έγγραφο, αλλά και να συλλάβω ουσιαστικέ παρατηρήσει για να συντάξω αυτό το έγγραφο. Μέχρι στιγμή έχω λάβει συγκεκριμένε προτάσει από τρει συναδέλφου και ένα email από τον κύριο Λούκε. Επομένω, συγγνώμη ξέχασα και τον κύριο Λόνε, τέσσερι συναδέλφου. Επομένω, αφού είναι κοινό το εγχείρημα αυτό, α εργαστούμε όλοι, α εργαστείτε και εσεί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είναι σημαντικό μετά από την έκκληση του, της συζυγήτριας για συνεισφορές όλοι να συνεισφέρουμε στη, στο έγγραφο εργασία. Ευχαριστώ τους διερμηνείς που μας χάρισαν λίγη ώρα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ξέρετε το χρονοδιάγραμμα, απόφαση 23-24 ε, Μαΐου, δημόσια κρόαση, εξέταση του σχέδιου έκθεσης πάει στις 29 Σεπτεμβρίου και περιμένουμε ε, συνεισφορές ε, από όλους στο έγγραφο εργασίας της εισηγήτριας. Ευχαριστώ όλους πολύ.